Bien. Nous allons ouvrir notre réunion. Je remercie mes chers collègues pour leur assiduité un lundi après-midi. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που είσαστε εδώ Δευτέρα το απόγευμα. Υιοθετούμε την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ούτε για τα πρακτικά. Τη συνεδριά του Δευτέρα Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις λοιπόν, θεωρούμε τα πρακτικά εγκεκριμένα. Τώρα στην ημερήσια διάταξή μας. Θέλαμε να η ανταλλαγή απόψεων. Θέμα η μελέτη που αναθέσαμε για την έμφυλη διάσταση στην πολιτική συνοχής. ο γενικός κανονισμός για το 2014-2020 για τα ταμεία μιλάει για την έλλειψη διάκρισης και ισότητα των φύλων και είναι μια οριζόντια αρχή για όλα τα ταμεία και αποτελεί προτεραιότητα όσον αφορά τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συχνά είναι δύσκολο για μας πραγματικά να λαμβάνουμε υπόψη τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχής, ΦΕΝΤΕΡ κλπ, τα διάφορα ταμεία, μπορούν στην πράξη να συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων με βάση το φύλλο. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να ανατεθεί μια ειδική μελέτη πάνω σε αυτό το θέμα. Και όπως υπενθύμησα στην προηγούμενη συνεδρίαση, αυτή η μελέτη ζητήθηκε από την απερχόμενη Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και παρεδόθη τον Φεβράριο 2019 η κυρία Μανουέλα Σαμέκ Λουντοβίτσι διεξήγαγε τη μελέτη από το Ινστιτούτο για τις Κοινωνικές Έρευνες με έδρα το Μιλάνο. Την ευχαριστώ πολύ που είναι παρούσα μεταξύ μας σήμερα το απόγευμα. Αυτή η μελέτη αναλύει λεπτομερώς το πώ η διάσταση των φύλων και η ισότητα ανδρών και γυναικών λαμβάνονται υπόψη στην πολιτική συνοχή στην περίοδο 2014-2020. Παρέχει στοιχεία με σκοπό τη βελτίωση της πρόθεση τη ισότητας των φύλων και της έλλειψης διάκριση μετά από το 2020. Είναι σημαντικότατο για μας να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε, κυρία μου, διότι διεξάγονται το διαπραγματεύσεις για τον νέο κανονισμό που θα ισχύει μέχρι το 2027. Αυτή η μελέτη έχει σκοπό επίσης να μας βοηθήσει να κάνουμε ένα απολογισμό της εφαρμογής αυτής της οριζόντιας αρχής. Να δούμε τι αποτελέσματα είχαμε, ποια θετικά αποτελέσματα, να καταλάβουμε τις αδυναμίες της υλοποίησης του προγράμματος. Είναι σημαντική συζήτηση, επίκαιρη, όλο και περισσότερο τα μάτια είναι πάνω μας, θέλουν να δουν πώς η αρχή της μη διάκρισης και η έμφυλη διάσταση λαμβάνονται υπόψη στις ευρωπαϊκές πολιτικές και πιο συγκεκριμένα στην πολιτική συνοχής. Με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν θα σας ακούσουμε. Και κυρία Λουντοβίτση σας δίνω το λόγο για 15 με 20 λεπτά. Μετά από αυτό θα διεξαχθεί συζήτηση που ελπίζω ότι θα είναι πολύ καλή συζήτηση και πλούσια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ήδη είπατε, αντικείμενο της μελέτης αυτής ήταν να αξιολογήσει το πώς ε, έχει γίνει ένα mainstreaming στην ε, διάσταση του φύλου για την προγραμματική περίοδο 14-20. τα βασικότερα ζητήματα ήταν πώς οι αρχές αυτές θα έχουν ενσωματωθεί σε όλα τα βήματα του κύκλου πολιτικής. Στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων. Υπάρχει λοιπόν πολύ υλικό που έχετε στη διάθεσή σας. Η έκθεση αυτή είναι το βασικό κείμενο. Μετά έχουμε παραρτήματα, πίνακες και όλες τις μελέτες περίπτωσης αυτό που κάναμε ήταν ότι υιοθετήσαμε την απλουστευμένη προσέγγιση ανάλυσης για την ε, διάσταση των φύλων, για το πώς θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την ισότητα των φύλων σε όλες σε τα πεδία παρέμβασης και τι πράγματι υλοποιήθηκε, που υπήρξαν αδυναμίες ή κενά στην εφαρμογή. προβήκαμε πρώτα μία ανάλυση της βιβλιογραφίας της εφιστάμενης, ε, επίσης ε, στατιστική μελέτη των ε, δεδομένων σχετικά με τις ενισχύσεις ή τα ποσά που διατίθενται και διεξήγαμε και μία έκθεση από φορείς, από μη καπαόμικρον, από υπηρεσίες που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων και τη διάστασή της σε διάφορα προγραμμάτα και κάναμε και 8 μελέτες περίπτωσης για κράτη, μέλη, επί τη βάση της κοινωνικο-οικονομικής τους κατάστασης και της κατάστασης της ισότητας των φύλων. Προσπαθώντας να έχουμε ένα διαφορετικό φάσμα ανάλογα προς τα κονδύλια που χρησιμοποιούν και ανάλογα προς την εδαφική κάλυψη. Επιλέξαμε Γερμανία και Γαλλία ως αρκετά αντιπροσωπευτικέ ε, των υπηρετικών, Ιταλία και Ισπανία ω αντιπροσωπευτικέ των νοτίων χωρών, Πολωνία και Ρουμανία ω αντιπροσωπευτικέ των ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών, την Ιρλανδία των αγγλοσαξονικών χωρών και τη Σουηδία των σκανδιναβικών χωρών, λέει ο Μιλήτρια. Και εδώ έχουμε μια, έναν κατάλογο των οκτώ λοιπόν μελετών περίπτωσης οι οποίες διατίθενται. Προτού πάμε στα όσα έχουν γίνει, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι στην ε, υφιστάμενη περίοδο προγραμματισμού, 14-20, υπάρχει μια αρκετά σημαντική ρυθμιστική υποστήριξη, όχι μόνο το άρθρο 7 των κοινών διατάξεων. Υπάρχει μια νομική βάση λοιπόν για το mainstreaming των φύλων, αλλά και άλλες προϋποθέσεις στον κανονισμό. Υπάρχει μια αιρεσιμότητα ex ante, που απαιτεί από τις χώρες να έχουν μια ικανή διοικητική ικανότητα και στρατηγικές, ώστε να υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων και στα θέματα πολιτικής συνοχής. Η αξιολόγηση εξάνεται εκτιμά τις δράσεις, τα μέτρα που έχουν τεθεί. Οι σχετικές υπηρεσίες και φορείς και μη καπαόμικρον θα πρέπει να συμμετέχουν στις εταιρικές αυτές σχέσεις και τις επιτροπές παρακολούθησης και οι αρχές διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμόζουν κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας που να μην είναι διακριτικής φύσεως και που να λαμβάνουν υπόψη τους την ε, διάσταση των φύλων και θα πρέπει να έχουν και ένα σύστημα παρακολούθησης με διαίρεση αναφύλο όπου δυνατόν και γιατί αιτήσει εκθέσεις επίσης πρέπει να παρουσιάζουν τα στοιχεία της υλοποίησης σχετικά με το πεδίο αυτό. Αυτό για όλα τα ταμεία. Από εκεί πέρα το κοινωνικό ταμείο έχει ιδιαίτερες ε, διατάξεις και υιοθετεί μια διτή προσέγγιση πέραν του mainstreaming των φύλων έχει και άλλα συγκεκριμένα μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τη σταδιοδρομία, την ισότητα, την μισθολογική και τη συμφιλίωση. Υπάρχουν όμως και κοινά, λέει ο Μιλήτρια. Υπάρχουν και κάποια κοινά. Ιδιαίτερα μια έλλειψη συγκεκριμένων θεματικών στόχων στα λοιπά μια πλην του κοινωνικού και αυτή η διτή προσέγγιση στα επιχειρησιακά προγράμματα αφήνεται στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Είναι λοιπόν εθελοντική και όχι υποχρεωτική προσθέτει ομιλήτρια και δεν υπάρχει συγκεκριμένη προϋπόθεση για όλα τα ταμεία να έχουν στατιστικές αναλύσεις αναφύλλω ή δυνατόν, αλλά τουλάχιστον επαρκείς δίκτες για τα φύλλα για παρεμβάσεις ε, υπό τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνολικά, η πολιτική συνοχής έχει υψηλές δυνατότητες στην υποστήριξη Τη ισότητα των φύλων και οι δυνατότητε αυτές δεν σχετίζονται μόνο με το κοινωνικό ταμείο αλλά και με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο συνοχή, τα οποία μπορούν να υποστηρίζουν σημαντικές δράσεις υπέρ τη ισότητα των φύλων, για παράδειγμα τα κενά στο πεδίο της έρευνας, γιατί υπάρχουν κενά στη σύνθεση των ερευνητών, Υπάρχει διαίρεση ανάλογα με τον ερευνητικό τομέα, αλλά και η έρευνα σχετικά με τις, διαφορές, με τις διαφορές των φύλων σε άλλα πεδία, λέει η ομιλήτρια. Το περιφερειακής ανάπτυξης έχει και μέσα εκτίμηση των δικτύων μεταφοράς και των, ε, της ε, Τεχνολογία της πληροφορίας, γιατί υπάρχουν διαφορές στο πώς τα φύλλα χρησιμοποιούν αυτά τα δίκτυα και επομένως στο σχεδιασμό των υποδομών αυτών πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές αυτές. Για τις νέες επιχειρήσεις, όπως και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχει μεγάλη διαφορά επιχειρηματικότητας μεταξύ των φύλων και εδώ το ERDF θα μπορούσε, θα μπορούσε να υποστηρίζει μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών στις startup εταιρείες στη νέα επιχειρηματικότητα αλλά και σε διευθυντικές θέσεις των επιχειρήσεων. Άλλες περιοχές τις οποίες το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να κάνει πολλά είναι στην υποστήριξη των κοινωνικών υποδομών και των κοινωνικών επιχειρήσεων για τη φροντίδα των ανηλίκων, των υπερηλίκων κτλ. Επομένως, χρησιμοποιώντα μια προσέγγιση συγκεκριμένη στα φύλλα, είναι δυνατόν να πετύχουμε πολλά. Και ε, αυτό ισχύει και για το ERDF, που φαίνεται να είναι ουδέτερο, λέει η ομιλήτρια, αλλά δεν είναι. Για να δούμε λοιπόν τις δυνατότητες των ταμείων αυτών σχετικά με την ισότητα των φύλων, κατηγοριοποιούμε όλες τις επενδυτικές ομάδες, κατηγορίες, 123 είναι επενδυτικές, και αυτές λοιπόν τις ταξινομούμε αναλόγως προς τη δυνατότητά τους για άμεση ή έμεση επίπτωση επί Τη ισότητα των φύλων. Και ταξινομώντας λοιπόν αυτές τι παρεμβάσει και βλέποντας τα συνολικά κονδύλια στο Open Cohesion Dataset περί το 57% των συνολικών προβλεπομένων για την πολιτική συνοχή κονδυλίων άμεσα ή έμεσα μπορούν να υποστηρίξουν την ισότητα των φύλων. Δυνητικά μπορούν Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τα μεγέθη αυτά στη διαφάνεια, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των ποσών αυτών είναι στο ESF, το 92%, αλλά και στο περιφερειακή ανάπτυξη έχουμε περί το 55% αν ακούσαμε καλά την ομιλήτρια, από τα κονδύλια δηλαδή που μπορούν δυνητικά και έμεσα να υποστηρίξουν τη ζωή των φίλων. Υπάρχει λοιπόν υψηλές, ε, υψηλό δυναμικό, υψηλές, ε, υψηλό περιθώριο δυνατοτήτων και αν δούμε αυτά τα στοιχεία αναχώρα, στα δεξιά, βλέπουμε ότι οι χώρες που έχουν υψηλότερες πιστώσεις σε αυτές τις ε, παρεμβάσεις, σε αυτού του είδους παρεμβάσεις, είναι οι σκανδιναβικές η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία ενώ αυτές που λιγότερο αφιερώνουν κονδύλια για τέτοιες παρεμβάσεις είναι οι ανατολικές χώρες με τη Ρουμανία να είναι ουραγός. Βλέποντας τώρα τις πιστώσεις για μέσα που άμεσα αφορούν στην ισότητα των φύλων. Αυτά τα λέμε 105, 105, είναι για την υποστήριξη ιδιαίτερα των θέσεων απασχόλησης για τις γυναίκες. 12 μόνον χώρες έχουν δεδομένα για τα κονδύλια εδώ. Και η Πολωνία φαίνεται να έχει το υψηλότερο ποσοστό εκατομμύρια ευρώ που έχουν επενδυθεί σε μέτρα άμεση στήριξη τη ισότητα των φίλων. Αν δούμε το μερίδιο των πιστώσεων αυτών ως προς το σύνολο και ιδιαίτερα στο ESF που έχει σημαντικές πιστώσεις για τέτοια μέτρα, μιλούμε για 2,5 μόνο περίπου τσεκατό για το σύνολο του ΕΣΕΦ. Με υψηλότερο μέρισμα στην Τσεχία, την Αυστρία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία. Άλλος ένας δείκτης που τον βρίσκει κανείς Καταρχάς να πω εδώ ότι έχουμε πολύ περιορισμένο υλικό, τουλάχιστον το 2018 είχαμε πολύ λίγο όταν διεξήγαμε την έρευνα προκειμένου να εκτιμήσει κανείς την διαφορά των φύλων στην κατανομή των πόρων, αριθμούς δικαιούχων κτλ. Ο μόνος κοινό δείκτης που μπορούσαμε να βρούμε ήταν ο αριθμός των έργων που υποστηρίζουν τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά απασχόλησης. Και κοιτώντας αυτά τα δεδομένα, ήταν σχετικά με την περίοδο 15-16 και είχαμε 5.694 έργα με το σκοπό αυτό, της υποστήριξης δηλαδή των γυναικών στην απασχόληση και της καταπολέμησης ε, των στερεοτύπων σχετικά με τα φύλλα. Τα δύο τρίτα των έργων αυτών υποστήριζαν τις θέσεις απασχόληση. 22% για κοινωνική συμπερίληψη και άλλο ένα σημαντικό ποσοστό για ε, επαγγελματική κατάρτιση. Και εδώ μιλούμε σε συντριπτική πλειοψηφία κονδύλια του ESF. Άνω των μισών εκ των οποίων υλοποιήθηκαν στην Γερμανία. Αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις κατανομές, τις πιστώσεις, τα έργα. Δεν έχουμε και πολλά στοιχεία. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη στις 8 χώρες που είχαμε επιλέξει. Και είδαμε τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης επιλέξαμε 28 επιχειρησιακά προγράμματα στις 8 αυτές χώρες για να δούμε τι ακριβώς συνέβαινε. Και αυτό που προέκυψε είναι ότι η συμφωνία αυτή της σύμπραξης εταιρικέ σχέσεις στις χώρες αυτές έχουν ισχυρή συνεκτίμηση της ισότητας των των φίλων ε, υπάρχουν γενικής, γενικές διακηρύξεις που λένε ότι η ισότητα των φύλων είναι πολύ σημαντική, ότι στα πλαίσια των ε, συμφωνιών αυτών πρέπει να γίνει ό,τι δυνατόν ώστε να υποστηριχθεί η ισότητα των φύλων, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με το πώς πρέπει να υλοποιηθεί μια τέτοια αρχή. Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς να διοργανώσει διαδικασίες επιλογής που να εφαρμόζουν αρχές αυτές, πώς να υποστηρίξει φορείς υπέρ της ισότητας των φύλων ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών. Δηλαδή πολλές δηλώσεις, αλλά πολύ λίγες ε, σαφείς ε, ενδείξεις στοιχεία για την υλοποίηση της προσέγγισης. Και αν δούμε τα επιχειρησιακά προγράμματα, στην ανάλυση πλαισίου υπάρχει πάντα η συμπερίληψη της αρχής της όντως των φύλων, αλλά στην υλοποίηση και πάλι πολύ λίγα πράγματα. Ιδιαιτέρως, εξετάζοντας το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο Κοινωνικό Ταμείο υπάρχει προτεραιότητα θεματικής παρέμβασης αλλά στο περιφερειακή ανάπτυξη δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Έχουμε λοιπόν σημαντικέ διαφορέ μεταξύ των χωρών, αλλά θετικό είναι ότι και οι οκτώ χώρες σημειώνουν μία βελτίωση στην παρούσα προγραμματική περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη και πολλές από αυτές έχουν αναπτύξει συγκεκριμένα εργαλεία υποστήριξης του mainstreaming των φίλων της ε, στην παρακολούθηση των έργων συνοχής. Δηλαδή φορείς συντονισμού που παρακολουθούν την υλοποίηση των ε, επιχειρησιακών προγραμμάτων και των εταιρικών συμφωνιών με ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα υπέρ της ισότητας των φίλων, Έχουν αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές και για τις αρχές ε, διαχείρισης και για τους δικαιούχους των έργων, προκειμένου να είναι αυτά πιο αποτελεσματικά στην υλοποίηση της αρχής της ισότητας των φύλων και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αναπτύξει και μέτρα βελτίωσης, αύξησης της ευαισθητοποίησης ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες, διότι εδώ χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δυνατότητες για να έχουμε καλύτερη ενσωμάτωση στην υλοποίηση της έννοιας της ισότητας των φίλων. Εδώ μπορείτε να δείτε τις επιστώσεις με τις ταξινομίες που σας έλεγα νωρίτερα. Πώς λοιπόν στις 8 αυτές χώρες τα κονδύλια σχετίζονται, μάλλον τα κονδύλια που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με την ισότητα των φύλων έχουν υλοποιηθεί. Και βλέπουμε ότι έξι χώρες έχουν μια συμμετοχή υψηλότερη από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 55%. Σε Ιρλανδία, Σουηδία, ε, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, αν ακούσαμε καλά. Για μέτρα άμεσα ή έμεσα, οι πιστώσει είναι πολύ υψηλότερε, αλλά είναι χαμηλότερε σε Πολωνία και Ρουμανία από τον μέσω όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δεν έχω διαφάνεια σε αυτό, αλλά ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα καλών πρακτικών. Στην ε, υλοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με μονομένα και κατακαιρματισμένα παραδείγματα, αλλά που μας δείχνουν ότι μπορούμε και με αυτό το Ταμείο κάτι να κάνουμε. Για παράδειγμα στη Γαλλία υποστήριξαν στις μεταφορές και τα διοργανωτικά για τα συνδικάτα των, ε, στον τομέα των μεταφορών την βελτίωση της συμμετοχής της ιότητας των φύλων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης. στην Ισπανία έχουμε πολλά προγράμματα υπέρ των νέων επιχειρήσεων και της γυναικείας επιχειρηματικότητας υπό το εμπορικά επιμελητήρια σε όλη τη χώρα, στη Σουηδία. Έχουν μέτρα ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής κατάρτισης στην δασοκομεία. Στην Ιταλία έχουν περιφερειακές συμφωνίες σύμπραξης μεταξύ επιχειρήσεων, κοινωνικών φορέων, ε, επιμελητηρίων και λοιπόν φορέων σε τοπικό επίπεδο, ώστε να υποστηρίζεται η γυναικεία απασχολησιμότητα, απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, ώστε να συμμετέχουν και οι επιχειρήσεις, οι ιδιωτικές και όχι μόνο οι δημόσιοι και λοιποί κρατικοί φορείς. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, αντίληψη από την πλευρά των ενδιαφερομένων φορέων, όπως σας είπα, κάναμε ε, ένα, ε, μια σφιγμομέτρηση και λάβαμε 42 απαντήσεις από διαφορετικούς δηλαδή οργανισμούς, ε, θεσμικά όργανα και μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις ε, και μετά μια δεύτερη με 23 συμμετέχοντες. Ε, και τι τονίστηκε εκεί. Τονίστηκαν ακριβώς τα ε, ισχυρότερα σημεία, αν θέλετε, αλλά και οι δυναμίε αυτών των προγραμμάτων σε ό,τι αφορά την διάσταση ακριβώς της ισότητα των φύλων. Σε ό,τι αφορά τα ισχυρότερα σημεία, είναι ακριβώς η εστίαση στη διάσταση του φύλου αλλά και η πολύ καλή νομική βάση με το άρθρο δηλαδή 7 του κανονισμού των κοινών διατάξεων και επίσης ε, το γεγονός ότι δίνεται ολοένα και περισσότερη πρόσοχη στη διάσταση του φύλου ε, στην εφαρμογή των διαφορετικών περιφερειακών πολιτικών στα διάφορα κράτη-μέλη και επίσης είναι θετικό το ότι αναπτύχθηκαν πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές και εργαλεία. Επίσης αναφέρεται ότι εκ των προτέρων ε, ρεσιμότητες, τα εξάντε conditionalities και οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις εξάντε evaluation σε ό,τι αφορά αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα και τη διάσταση του φύλου αποτέλεσαν πολύ σημαντικά εργαλεία προκειμένου να υπάρξει περισσότερη ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά τη μειοθέτηση αυτής της διάστασης. Όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και σε άλλα ταμεία. Ποια είναι τώρα τα κυριότερα, οι κυριότερες αδυναμίες, αν θέλετε. Πάλι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα σε ό,τι αφορά αφενός τον προγραμματισμό και αφετέρου την εφαρμογή, την υλοποίηση. Δηλαδή, ε, συχνά θεωρείται πως η διάσταση του φύλου αποτελεί ένα οριζόντιο, ε, μια οριζόντια γενική διάσταση, αλλά δεν υπάρχει ε, πιο συγκεκριμένη εφαρμογή. Δηλαδή δεν υπάρχει αντίληψη του γεγονότος ότι η λήψη υπόψη της διάστασης του φύλου είναι σημαντικότατη για την οικονομική ανάπτυξη. Όχι μόνο δηλαδή σημαντική για τις κοινωνικές αξίες και ούτω καθεξής, αλλά και για την ίδια την οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλές δηλαδή μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν ότι οι χώρες εκείνες οι οποίες έχουν περισσότερη ισότητα των φύλων σε όλε τι διαστάσει τη οικονομική ζωή, επιτυχάουν ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη από ό,τι άλλε χώρε σε Ένα άλλο πρόβλημα είναι η ελλείψη ευαισθητοποίηση, η αντίληψη αυτού του ζητήματο. Και αυτό αναφέρεται από του διάφορου αρμόδιου φορεί, του stakeholders δηλαδή, πολλέ φορέ και αρμόδιε διοικητικέ αρχέ, αλλά και όσοι εποφελούνται από αυτά τα project δεν γνωρίζουν, δεν έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και δεν έχουν απαραίτητη κατάρτιση ούτως ώστε να γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν αυτή τη διάσταση του φύλου. Και ένα ακόμα ζήτημα το οποίο ε, προέκυψε είναι η έλλειψη πολιτικής δέσμευσης. Δηλαδή το ζήτημα της διάστασης του φύλου λαμβάνει λιγότερη ε, προσοχή σε, όλες τις, ε, σε όλους τους ομίσους πολιτικής κατά τελευταία χρόνια. Αυτά και περνάω τώρα στα συμπεράσματα και στα διδάγματα που αντλήσαμε με βάση τα όσα προέκυψαν και αυτό που μπορούμε να πούμε περιληπτικά είναι ότι η πολιτική συνοχή μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την προώθηση τη διάσταση ακριβώ τη ισότητα των φύλων σε μία σειρά από τομεί παρέμβαση. Μπορεί να υποστηρίξει δηλαδή τη λήψη άμεσων μέτρων στου διάφορου τομεί ε, παρέμβαση, στι διάφορε περιοχέ παρέμβαση, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα υπόδειγμα και μια κινητήριο δύναμη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή περιφερειακών πολιτικών από τα κράτη-μέλη στον τομέα τη διάσταση του φύλου. Και το έχουμε δει να λαμβάνει ε, χώρα ε, στην πράξη, ότι δηλαδή οι εθνικέ αλλά και περιφερειακέ πολιτικέ μπορούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάπτυξη των δικών του ε, πολιτικών. Αλλά υπάρχουν και τα προβλήματα που ήδη Αναφέρθηκαν δηλαδή το χάσμα ανάμεσα στον προγραμματισμό και την εφαρμογή, η ελλειπής γνώση και η ελλειπής ε, τεχνογνωσία των εισαγωγικών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτής της διάστασης του φίλου στην πράξη ε, και επίσης αδυναμία σε ό,τι αφορά τον, ε, τον σχεδιασμό των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων αλλά και η έλλειψη πολιτικής δέσμευσης. Σε ό,τι αφορά τώρα την πολιτική συνοχής μετά από το 2020 με βάση το ερωτηματολόγιο και τι απαντήσει που λάβαμε από του stakeholders, του συναρμόδιου εφορεί, υπάρχει σκεπτικισμό σε ό,τι αφορά το πώ η νέα προγραμματική περίοδο ε, θα αλλάξει την υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό δηλαδή που ανέφεραν είναι ότι ε, δίνεται λιγότερη προσοχή στο ζήτημα της διάστασης του φύλου, τουλάχιστον στο σχέδιο του κανονισμού που προετοιμαζόταν πέρυσι. Δηλαδή δεν δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση ε, στα ζητήματα της διάστασης του φύλου, της ισότητας ε, των φύλων. Και αυτό τι σημαίνει με τη σειρά του, ότι αντίστοιχα δίνεται λιγότερη προσοχή σε ό,τι αφορά τη λήψη υπόψη της διάστασης της ισότητας των φύλων και στο εθνικό και στο περιφερειακό επίπεδο. Άρα λοιπόν υπάρχει ε, φόβος ότι στη νέα προγραμματική περίοδο θα υπάρξει ασθενέστερη υποστήριξη της ε, διάσταση ε, τη ισότητα των φύλων. Άρα λοιπόν, ποιες συμπερασματικά είναι οι συστάσει μα ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η εστίαση σε αυτό το ζήτημα και θα πρέπει επίση να παρασχεθεί συγκεκριμένη υποστήριξη και κατευθυντήρε γραμμέ έτσι ώστε να μπορούμε να ε, εφαρμόζουμε αυτή την διτή, αν θέλετε, προσέγγιση. Όχι λοιπόν μόνο κατεύθυνση και κατευθυντήρε γραμμέ, καθοδήγηση δηλαδή, αλλά και συγκεκριμένα εργαλεία για την εφαρμογή αυτή τη διάσταση. Ε, θα πρέπει δηλαδή να διατηρηθεί ο στόχος της διάστασης του φύλου σε όλα τα ταμεία για την περίοδο μετά το 2020 και επίσης θα πρέπει να εφαρμοστεί η συμμόρφωση με τα ζητήματα του φύλου, για παράδειγμα, με με την επιβολή υποχρεωτικών δεσμευτικών προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά την ε, διάσταση του φύλου, σε ό,τι αφορά και την επιλογή των ε, επιλέξιμων ε, project αλλά και την αξιολόγησή τους. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερη παράδοση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτής της διάστασης, ο στόχος είναι να βελτιωθεί η ικανότητα προς αυτή την κατεύθυνση όλων των ε, αρμοδιών ε, φορέων μέσω ε, και της κατάλληλης πολιτικής καθοδήγησης αλλά και μέσω συγκεκριμένων εργαλείων. Ένα παράδειγμα για παράδειγμα είναι αυτό της Ισπανίας όπου δημιουργήθηκε αυτό το δίκτυο στα ταμεία συνοχής για τη διάσταση του φύλου και το οποίο δίκτυο ήταν πολύ αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά ακριβώς την προώθηση της περισσότερες υψηλότερες ευαισθητοποίησεις σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη, την λήψη υπόψη της διάστασης του φύλου στις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές. Επίσης, εκείνο που λέει σημαντικό είναι ότι το γεγονός ότι θα πρέπει να ληφθεί καλύτερα υπόψη αυτή η διάσταση και ε, στο επίπεδο των ε, αρχών τοπική και περιφερειακή ε, αυτοδιοίκηση, δηλαδή όχι μόνο θεωρητικά, αλλά πραγματικά να συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι αφορά τη χάραξη των σχετικών πολιτικών και επίσης θα πρέπει να υπάρξουν στοιχεία δεσμευτικά της διάστασης του φύλου τα οποία θα επιβάλλουν την συμπερίληψη δικτών που θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση αυτοί. Δηλαδή, όχι μόνο δείκτε οι οποίοι, για παράδειγμα, θα αφορούν μόνο τα δύο διαφορετικά φύλλα, αλλά και δείκτε σε ό,τι αφορά το τι ακριβώ λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο του προγράμματο για τη διασφάλιση τη ισότητα των φύλων. Και επίση θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη πολιτική δέσμευση τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε εθνικό επίπεδο. Θα σταματήσω εδώ. Ελπίζω να ήμουν ασαφή και αν υπάρχουν ερωτήματα, είμαι στη διάθεσή σα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κυρία Λουντοβίτση για τις πληροφορίες αυτές. Υπήρξατε σαφέστατοι. Μας ενημερώσατε εδώ, όντως, μάθαμε πολλά σχετικά με τα εναπομένοντα να γίνουν προς επίτευξη των στόχων όσον αφορά τη μη διάκριση και πώς θα λάβουμε υπόψη την έμφυλη διάσταση. Αυτή η συζήτηση διεξάγεται την πιο κατάλληλη στιγμή στην Επιτροπή μας, διότι όπως σας είπα συζητούμε το θέμα αυτό. Σημείωσα την απεσιόδοξη νότα που εκφράσατε στο τέλος όσον αφορά το μελλοντικό προγραμματισμό, τουλάχιστον από την πλευρά των δικαιούχων. Εκφράσατε κάποιο φόβο κατά πόσο θα λαμβάνετε επαρκώς υπόψη αυτή η διάσταση. Ελπίζουμε να σας διαψεύσουμε, να διαψεύσουμε εκείνους που εκφράζουν φόβους σήμερα. Ε, βάσιμους φόβους, δυστυχώς. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο συνάδελφός μας, ο κ. Αϊμού, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε πολύ κυρία Λουντοβίτση για αυτή την ενδιαφέρουσα ανάλυση που ακούσαμε ε, και το υλικό το οποίο μας παρουσιάσατε. Βέβαια δεν διάβασα όλο αυτό το υλικό, αλλά σας άκουσα προσεκτικά και ε, ισχύει πράγματι ότι η ισότητα των φύλων Ε, δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε διαρκώς κατά νου όταν χαράζουμε τις πολιτικές μας ε, και γι' αυτό είναι καλό το ότι υπάρχουν τέτοιου είδους μελέτες οι οποίες μας υπενθυμίζουν ότι πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτή τη διάσταση. Επίσης ήταν ενδιαφέρον το, ε, το συμπέρασμα που αντλείτε με βάση την ανάλυση σας ότι τα νέα κείμενα τα οποία εκπονούνται αυτή την ε, περίοδο και ήδη προκατακτικέ εργασίε ε, που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίνονται στι προσδοκίε σα. Ότι δηλαδή η διάσταση τη ισότητα των φύλων δεν ε, λαμβάνεται αρκόντως, υπόψη. Και στη σελίδα 105 του εγγράφου σας διάβασα ένα συμπέρασμα το οποίο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτό και να μην αναφερθώ σε κάτι άλλο. Αναφέρεστε λοιπόν εκεί ότι υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα αφενός στην απλούστευση των ταμείων εύση και αφετέρου στη λήψη υπόψη της διάστασης της ισότητας των φύλων. Δηλαδή, προσπαθούμε από τη μία πλευρά να διαμορφώσουμε με πιο απλό τρόπο τα διάφορα αυτά τα ταμεία με αποτέλεσμα να δίνουμε ε, λιγότερη έμφαση στη διάσταση της ισότητας των φύλων. Αυτό τουλάχιστον μας λέτε εδώ συμπερασματικά. Ε, γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό και πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τους δύο στόχους αυτούς παράλληλα, δηλαδή και να δώσουμε περισσότερη έμφαση στη διάσταση του φύλου και από την άλλη να απλουστεύσουμε στη δομή του στα ταμεία έρευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε απευθείας στο ερώτημα του συναδέλφου μας, ούτω ώστε η συζήτηση να έχει μεγαλύτερο δυναμισμό. Ε, σας έχετε, έχετε το λόγο. Πράγματι, υπάρχει μια φαινομενική αντίφαση, διότι δεν υπάρχει επαρκής γνώση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ότας των φίλων σε όλα τα ταμεία. Όταν μαθαίνει κανείς βλέπει ότι δεν είναι τόσο δύσκολο, υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία, έχουν αναπτυχθεί επί σειρά ετών και μπορούμε να δούμε που υπάρχει ανάγκη για παρέμβαση. Πώς μπορούμε να παρέμβουμε, τι δείκτες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τι είδου εργαλεία εποπτικά, ποια κριτήρια και διαδικασία επιλογής. Το ότι απλούστευση σημαίνει περικοπή δεν είναι σωστή αντίληψη. Διότι τα ταμεία θα είναι λιγότερο αποτελεσματικά από ό,τι θα έπρεπε. Ήταν πολύ σημαντικά μέχρι το ισότητα των φύλων, κυρίω εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα σε χώρε. Δεν θεωρείτο σαν πρόβλημα η ισότητα των φύλων. Είναι κρίμα τελικά αν έχουμε απώλειες λόγω της ιδέας, της αντίληψης αυτής που υπάρχει περί απλούστευσης. Ευχαριστώ πολύ. Μόνικα Βένα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λουντοβίξη και τους συντάκτες, τους υπόλοιπους της έκθεσης. Έξοχη μελέτη, πολύ ενημερωτική, σαν πράσινη ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για αυτή τη μελέτη. Χαιρόμαστε που την έχουμε στα χέρια μας. Αυτή η Επιτροπή πραγματικά θα πρέπει να λάβει υπόψη σοβαρότατα τα πορίσματα και τις τάσεις της εκθέσεως, διότι έχουμε δουλειά μπροστά μας. Η διάσταση του φύλου είναι, θα έπρεπε να είναι κάτι προφανές και να εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα και στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη καταδεικνύει ότι στη φάση προγραμματισμού, στις συμφωνίες συνεργασίας και στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται υπάρχει διάστηση φύλου στην ε, υλοποίηση λείπει παντελώ. Κυρίω στο ERF, όχι στο ESF. Στο Περιφερειακό Ταμείο ε, περιφερειακή ανάπτυξη υπάρχουν ελλείψεις. Εμείς σαν πράσινοι θέλαμε ακριβώ αυτή τη μελέτη. Θέλαμε να θέσουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, Διότι δεν είναι προφανέ σε αυτά τα μία πώ θα εφαρμόσει τη διάσταση του φύλου. Και αυτό είναι και δουλειά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υποβάλει σχετικές προτάσεις. Και ο νέος αρμόδιος επίτροπος θα πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις με θέμα την εξασφάλιση της ε, εφαρμογής της διάστασης του φύλου στην πολιτική συνοχής. Σκεφτείτε ότι η πολιτική συνοχής είναι το σημαντικότερο επενδυτικό εργαλείο στη διάθεσή μας στην Ευρώπη. και για την εφαρμογή της διάστασης του φίλου Είναι πολύ σημαντικό μέσο. Ήδη είπατε ότι υπάρχουν δύο πυλώνες όσον αφορά δυνατότητες, στοχευμένη δράση και οριζόντιοι στόχοι. Πολύ δουλειά απομένει να γίνει. Από την εμπειρία μου ισχύει αυτό που είπατε. Οι εμπειρογνώμονες όταν συνομιλεί κανείς μαζί του, μαζί τους, λένε ότι ίσως θα πρέπει να φοβηθούμε και κάποια αρνητικά αποτελέσματα, κάποια αντίδραση και ε, η παναχώρηση σχέση με τα επιτευθέντα. Πρέπει να μας ξυπνήσει αυτή η, αυτή η έκθεση και η Επιτροπή μας να λάβει σοβαρότατα υπόψη το θέμα. Να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις. Κυρίως στις περιφέρειες και στις πόλεις πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο στόχος της διάστασης της ότες των φύλων στην ε, πολιτική συνοχής. Ένα από τα προβλήματα που ήδη δείξαμε και στις διαπραγματεύσεις για το CPR ήταν η βελτίωση των στοιχείων των, ε, που είναι, δεν είναι ομαδοποιημένα πλέον κατά αναφύλλο και στην Επιτροπή Γυναικών και στο φορέα την των φίλων το έθεσε αυτό. Και η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με την Επιτροπή Γυναικών να δούμε πώς θα έχουμε πιο λεπτομερή στοιχεία που θα λαμβάνουν υπόψη την πολιτική συνοχή. Αν δεν έχουμε αναφύλω στοιχεία, τα πράγματα περιπλέκονται για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συγκεκριμένα εργαλεία και προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Ήδη αναφερθήκατε σε κάποιες συστάσεις. Δεν θέλω να τις επαναλάβω. Χρειαζόμαστε σαφείς προσανατολισμούς, αυτό είναι που χρειαζόμαστε για τα εργαλεία που θα εφαρμόσουμε για την ισότητα των φύλων Χρειαζόμαστε και καθορισμό στρατηγικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. και να διατηρηθούν και τα εκ των προτέρων κριτήρια. Θα λάβουμε σοβαρότατα υπόψη μας τα κριτήρια αυτά. Θα τα επεξεργαστούμε και θα αυξήσουμε και τι πιέσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτω ώστε να παρουσιάσει ουσιαστικέ προτάσει για τη βελτίωση της καταστάσεω τάχιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ιζαμπέλ Μπενζαμέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίαση. ο πιο σημαντικός στόχος των ευρωπαϊκών ε, προγραμμάτων και έργων είναι να βελτιώσουν την πρόσβαση και των δύο φύλων ε, στις ε, ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά απασχόλησης. Και επομένως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ισότιμο παιχνίδι στην πρόσβαση αγοράς απασχόλησης. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα σε κάτι που είπατε για την γυναική επιχειρηματικότητα. Δηλαδή τον αριθμό των γυναικών πού ξεκινούν νεε επιχειρήσεις, πού συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και αναφερθήκατε σε μια σειρά από περιορισμούς σχετικά με την πρόσβαση στην πίστοση και σε άλλους περιορισμούς. Δηλαδή στην ανάπτυξη μιας νέα επιχειρηματική δραστηριότητας στην Ευρώπη. Πόσο σημαντικές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε που θέλουν να είναι επιχειρηματίε σε σχέση με άνδρε που βρίσκονται στην ίδια κοινωνική οικονομική κατάσταση, στην ίδια ηλικία, στην ίδια χώρα κτλ. Δηλαδή η πραγματική ποιοτική διαφορά μεταξύ των φίλων στη νέα επιχειρηματικότητα ποια ακριβώ είναι. Σα ευχαριστώ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Λουντοβίτσι ε, να, απαντήσει αν θέλει. Ε, κοιτάξτε δεν έχω τα δεδομένα αυτή τη στιγμή αλλά είχαμε μία μελέτη από το AG τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ισότητα των Φύλων, με μια εστίαση στη γυναική επιχειρηματικότητα και έχουμε πλέον αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι συνήθως οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περιορισμό πίστοσης, δηλαδή ε, δεν έχουν επαρκής, επαρκή κονδύλια πίστοσης στην επιχειρηματικότητα Επίσης υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των φύλων, ένας διαχωρισμός στο πώ δημιουργούνται οι επιχείρησει. και μετά υπάρχουν και τα διάφορα προβλήματα της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, διότι επιχειρηματικότητα σημαίνει ε, πολλές ώρες απασχόλησης, δύσκολο να το συνδυάσει αυτό κανεί με οικογενειακέ υποχρεώσει. Αλλά είδαμε και μία μελέτη του ΑΣΑ που δείχνει ότι και ο τρόπος, η προσέγγιση είναι διαφορετική μεταξύ των φίλων. Δηλαδή οι γυναίκες προσέχουν περισσότερο το μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδο δυνατότητας κερδοφορίας. Αποφεύγουν τον κίνδυνο περισσότερο, το ρίσκο, και αν θέλετε συμπληρώνουν την ανδρική επιχειρηματικότητα και παρέχουν μια πολύ καλή υποστήριξη τη δομή της οικονομίας, στα θεμέλια της οικονομίας. Όταν μιλούμε για την προσέγγιση γιούνους, την μικροπίστοση... η προσπάθεια εκεί είναι να συνεργαστούν με γυναίκες γιατί δεν τους ενδιαφέρει το υψηλό ρίσκο, τους ενδιαφέρει το μέσο μάκρο πρόθεσμο επίπεδο. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικές υπηρεσίες ο σχετικός τομέας των επιχειρήσεων αυτών και σε πρόσφατη βιβλιογραφία ε, ε, σημειώνεται η σημασία της γυναικείας επιχειρηματικότητας διότι διαφοροποιεί ή αν θέλετε εξισορροπεί την οικονομική δραστηριότητα και παρέχει νέες προσεγγίσεις ώστε οι επιχειρήσεις να επενδύουν με διαφορετικό τρόπο. Δημιουργεί, αν θέλετε, διαφορετικότητα, που και αυτή είναι σημαντική. Και υπάρχει και σε αυτή τη μελέτη λοιπόν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε. Στεφάν Μπιζού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση με το Renew. Τα τελευταία που είπατε δεν το ακούμε ως σύσταση αλλά ως σήμα κινδύνου. Δηλαδή αυτά που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη ε, σας φαίνονται επαρκώς ε, ευάλωτα ώστε ίσως να έχουμε υποχώρηση στα επόμενα χρόνια και αυτό μας θυμίζει το εξή. ότι η δουλειά που γίνεται επί της ισότητας των φύλων κρύβει την ισότητα ευκαιριών. Και εδώ αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλούς τομείς της συλλογική μας δραστηριότητας αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι ακόμα πιο ανησυχητικός όταν εμφανίζονται ακριβώς στο πόσο ισότιμες είναι οι ευκαιρίες για τα δύο φύλλα και αυτό ενισχύει την συλλογική μας ευθύνη να παρέμβουμε μέσω μέτρων συνοχής και θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και θα θέλαμε να μοιραστείτε τα στοιχεία και τους δείκτες που έχετε μαζί μας γιατί ε, θεωρούμε ότι συλλογικά από κοινού μπορούμε να μετακινήσουμε τα όρια αυτά ή τους περιορισμούς. Εσείς εξετάσατε ε, κάποιες περιπτώσεις στη μία ή στην άλλη χώρα κάποιο εκπληκτικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, ώστε να σκεφτείτε ότι αυτό θα έπρεπε να μοιραστούμε με τις υπόλοιπες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα καλό δηλαδή προς μίμηση παράδειγμα. Σας ευχαριστώ. Σας απαντήσει η κυρία Λοντοβίτσι. Ναι, πράγματι. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου γιατί δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το ζήτημα. Ειδικότερα με την κρίση ε, των τελευταίων χρόνων δεν είχε πλέον το ίδιο ειδικό βάρος η διάσταση του φύλου. Και βέβαια πρόκειται και ένα ζήτημα ε, πόρων, αν θέλετε. Γιατί βέβαια οι γυναίκες λαμβάνουν λιγότερη εκπαίδευση από τους άντρε, αλλά στη συνέχεια όταν κάνουμε προσπάθειες για να λάβουν περισσότερη εκπαίδευση, ουσιαστικά ε, κατασπαταλούμε αυτή την, την περισσότερη κατάρρευση που λαμβάνουν, γιατί δεν του δίνουμε τι απαραίτητε εργασιακέ ευκαιρίε και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά τώρα τι ε, βέλτιστε πρακτικέ, ε, στην ε, έκθεση αναφέρουμε κάποια παραδείγματα, ναι, πολύ ενδιαφέροντα δηλαδή παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, τα οποία ανέφερα ε, συνοπτικά προηγουμένως, ε, δηλαδή ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση του φύλου στους τομείς εκείνους οι οποίοι παραδοσιακά, αν θέλετε, δεν λαμβάνουν υπόψη αυτό το ζήτημα ή δεν ε, δίνουν την, την προτεραιότητα που χρειάζεται, για παράδειγμα, ο τομέας των μεταφορών, ο τομέας της δασοκομείας και ούτω καθεξής Και εδώ είναι σημαντικό να υπάρχουν αρμόδιοι φορεί οι οποίοι θα συντονίζουν την όλη προσπάθεια και θα την εποπτεύουν έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούν κατά την εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλίων τι ακριβώς λειτουργεί στην πράξη και τι όχι, έτσι ώστε να λαμβάνουν και τα συμπληρωματικά μέτρα και να βελτιώνουν την κατάσταση με την παροχή περαιτέρω κατάρτισης, με τεχνική αρρωγή, με την παροχή των απαραίτητων εργαλείων. Γιατί όπως είπα, ήδη έχουν, ε, έχουμε στη διάθεσή μας τα απαραίτητα εργαλεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό. Το πρόβλημα όμω είναι ότι συχνά σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο δεν υπάρχει γνώση αυτών των εργαλείων και του τι ακριβώ μπορεί δηλαδή να γίνει για να προωθηθεί η διάσταση του φίλου μέσω τη πολιτική συνοχή. Και ακριβώ εδώ θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη διάχυση αυτής της γνώσης, να υπάρξει περισσότερη γνώση ότι υφίστανται αυτά τα εργαλεία προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή αυτή τη διάσταση στι πολιτικέ. Δηλαδή δεν θα πρέπει να δοθεί εσφαλμένη εντύπωση ότι τα έχουμε κάνει ήδη όλα και δεν χρειάζεται πλέον να επενδύσουμε περισσότερο σε αυτό. Όχι, θα πρέπει να συνεχιστούν οι επενδύσεις. Ε, και η μελέτη των εμπειρογνωμόνων από τη Σουηδία αναφέρει, και μάλιστα στη Σουηδία εκεί μιλάμε για πολύ ανεπτυγμένη λήψη υπόψη τη διάσταση του φύλου. Αναφέρει λοιπόν εκείνη η μελέτη ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια που γίνεται σε ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα του δικαιούχου ε, των διαφόρων ε, προγραμμάτων, ειδικότερα στο ε, Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και ούτω καθεξή. Δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Ευχαριστώ πολύ την κυρία ε, Λοντοβίτσι για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Θα ξεκινήσω με μια παρατήρηση από την πλευρά μου. δηλαδή, ε, δίνεται ε, συχνά η εντύπωση ότι έχουμε κάποια κονδύλια τα οποία κατευθύνονται για παράδειγμα για τη διάσταση του φύλου ή όχι, ουσιαστικά δηλαδή δεν υπάρχουν κονδύλια αν θέλετε ουδέτερα, τα οποία δηλαδή δεν αφορούν αν θέλετε αμύγό σε άντρες ή γυναίκες ή οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτό χρειάζεται αυτό να υπάρχει και στο επίπεδο της υποδομής. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό σε επίπεδο υποδομής όταν κάνουμε για παράδειγμα μία, όταν κατασκευάζουμε αυτοκινητόδρομο ή κατασκευάζουμε για παράδειγμα μία σιδηροδρομική ε, τροχιά. Γιατί για παράδειγμα, όταν λέμε ότι κατασκευάζουμε αυτοκινητόδρομο, υπάρχει για παράδειγμα κυβερνητικό σταθμό κατά μήκο, μπορεί να διευκολυνθεί δηλαδή ε, περισσότερο η γυναίκα. Όλα αυτά λοιπόν λαμβάνονται, παραδειγμα βρεφονικο σταθμο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ε, τώρα, στην Ανατολική Γερμανία και ιδιότερα στις αγροτικές περιοχές έχουμε μεν μεγάλη μετανάστευση από αυτές τις ε, περιοχές προς ε, άλλες περιοχές της της Γερμανίας αλλά δεν παρατηρείται τόσο έντονα αυτό το φαινόμενο σε ό,τι αφορά τις γυναίκες που έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε αυτές τις γυναίκες να παραμείνουν εκεί σε αυτές τις περιοχές. Θεωρείτε ότι υπάρχει ε, ε, ε, κάτι τέτοιο, ένα φαινόμενο αντίστοιχο το οποίο παρατηρείται και αλλού, το ότι δηλαδή ε, ασκείται ιδιαίτερη πίεση λόγω των περιστάσεων στις γυναίκες με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους. Μετά, αναφερθήκατε στο κείμενο του κανονισμού και το γεγονός ότι κατά την άποψή σας δεν ε, λαμβάνεται παρκώς η διάσταση του φύλου εκεί. Τι ακριβώς δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να γίνει παραπάνω. Και πράγματι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε ότι θα πρέπει να διαδώσουμε περισσότερο το, αυτό το ζήτημα και να το λαμβάνουμε ε, υπόψη μας και αυτό σημαίνει βέβαια ότι και οι διάφοροι επίτροποι θα πρέπει να ε, έχουν πάντοτε κατά αυτή τη διάσταση του φίλου Δηλαδή και οι πολιτικοί θύνοντες των ε, αρχηγοί των κρατών ε, μελών ε, και των ε, κυβερνήσεων αλλά και οι, επίτροποι θα πρέπει να κάνουν μια ε, συντονισμένη προσπάθεια και ενδεχομένω θα πρέπει να δημιουργηθούν και οι απαραίτητε συμμαχίε, όπω για παράδειγμα αυτό το δίκτυο το οποίο αναφέρατε στην Ισπανία το, οι οποίοι ακριβώ μπορούν να ενισχύσουν ακριβώ τη λήψη υπόψη τη διάσταση τη ισότητα των φύλων. Και επίση, εκείνο που χρειαζόμαστε απαραίτητα είναι να υπάρχει και η απαραίτητη παρακολούθηση και επίσης ε, να έχουμε και τα δεδομένα τα οποία θα συγκεντρώνονται και σε επίπεδο φίλων, ώστε να γνωρίζουμε πώ ακριβώ δαπανούνται τα κονδύλια μα. Δηλαδή, είναι μεγάλο κρίμα ε, το γεγονό ότι δαπανούμε κονδύλια σε ό,τι αφορά τη συμμετοχική οικονομική ανάπτυξη ε, και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή που δεν επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον και δεν αυξάνει τι ε, εκπομπέ άνθρακα. Άρα λοιπόν, αφού κάνουμε αυτή την προσπάθεια, πρέπει να αξιοποιήσουμε τη φάση μετάβασης και μετάλλαξη ε, που διέρχεται η οικονομία μας σε ό,τι αφορά ακριβώ τη λήψη υπόψη των περιβαλλοντικών και άλλων ζητημάτων. Εάν λοιπόν θέλουμε να εφαρμόσουμε ορθά την νέα οικονομική μα ανάπτυξη, το νέο μοντέλο, τότε θα πρέπει να λάβουμε αρκούντω υπόψη και αυτή τη διάσταση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκοπούν από αυτή την οικονομική ανάπτυξη οι ασθενέστερε οικονομικά περιοχέ. Ευχαριστώ πολύ, Ρόζα Νταμάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την σιγήτη για τη μελέτη. Δύο ερωτήσει έχω καταρχήν. Έριξα μια ματιά και στα διάφορα παρατημάτα και είχα την εντύπωση ότι η χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι το πιο ενδεδειγμένο, η πιο ενδεδειγμένη λύση. Διότι πιστεύω ότι η γυναίκα χρειάζεται περισσότερο να βρει δουλειά και να την κρατήσει μετά. και για να μπορεί να χειριστεί την κατάσταση στην οικογένεια με τους ηλικιωμένους και τα παιδιά. Το βλέπουμε αυτό σε κράτη-μέλη όπου υπάρχει πρόνοια. Που να μελετήσουν, είναι πιο εύκολο να μελετούν τα παιδιά και το απόγευμα. Δεν υπάρχει αυτό στα κράτη-μέλη όπου τελειώνει το σχολείο το μεσημέρι. Λοιπόν, μίσο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι πιο δεδειγμένο για βοηθήσει τη γυναίκα να αντιμετωπίσει αυτού του είδου τα προβλήματα. Και εγώ θα ήθελα ομαδοποιημένα στοιχεία. αναφύλων ή θέλαμε να ξέρουμε ποιες θέσεις εργασίας βοήθησε το Ταμείο Συνοχής να δημιουργηθούν, σε ποια κοινωνικά στρώματα, για την καταπολέμηση της φτώχειας. Η βοήθεια να δουλέψει γυναίκα είναι κάτι σημαντικό. Θέλουμε να δούμε σε ποιο βαθμό. Και κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τη διαφορά της οικονομικής αντιμετώπισης που υπάρχει μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη και τι μπορεί να κάνει και για αυτό το θέμα η πολιτική της ε, συνοχής. Απάντηση, ναι. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι πιο εύχριστο για θέματα ισότητας των φύλων. Προωθεί την κοινωνική συμπεριλήψη, απασχόληση, κατάρτιση, παιδεία, στοχευμένα μέτρα σε ατομικό επίπεδο είναι ένα πολύ σημαντικό ταμείο, κρίσιμη σημασία του για την ιστότητα των φύλων. Και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και αυτό μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, να υποστηρίξει την έρευνα, κάποια είδη έρευνας, τους ερευνητές και στοιχεία αναφύλου θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμα υποστήριξη πολιτικών μεταφοράς πληροφορικής για να βοηθήσουμε όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν περισσότερες δημόσιες μεταφορές από τους άντρες. Σε διαφορετικές ώρες και χρειάζεται να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στις μεταφορές γιατί έχουν και μέλη της οικογένειας. Χρειάζονται φωτισμό, καλό, ασφάλεια κλπ. Αυτή η τομή πολιτικής είναι σημαντική και για την ισότητα των φύλων και μέχρι τώρα δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς. Είναι λιγότερο αναπτυγμένοι οι Όσον αφορά την ισορροπία οικογενειακή ε, ζωής και εργασία. αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για τις γυναίκες, αλλά όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρες. Εκείνους που πρέπει να φροντίσουν γονείς, παιδιά, αληθεύει ότι πρέπει να μην πούμε ότι χρειάζεται μόνο η δομή, υποδομή φροντίδας, αλλά τι ώρα είναι ανοιχτά, τα, ανοιχτές οι διαφορές υπηρεσίες. Ε, όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζονται αυτού του είδους υπηρεσίες. Αναφερθήκατε και στην Ήπεθρο. Κάναμε μία μελέτη συναθρήσαμε την ισότητα των φύλων με τη δημογραφική αλλαγή. Είναι αλληλένδετα θέματα. Ο γυρεότερος πληθυσμός αποτελείται κυρίως από γυναίκες που ζουν μόνες τους. Πολύ συχνά στην ύπεθρο και χρειάζονται κάποια υποστήριξη. Πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Εάν δούμε ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή, πρέπει να βρούμε κατάλληλο μέτρο, να βρούμε απάντηση να μην λέμε αόριστα θέλουμε ισότητα των φύλων. Εδώ η ισότητα των φύλων έχει ιδιαιτερότητες και χρειάζεται ειδική παρέμβαση. Ποια είναι η ιδέα. Πάντα να φοράμε τα γυαλιά αυτά της ισότητας των φύλων. Βλέποντας μέσα από αυτά βρίσκεις λύσεις που διαφορετικά δεν θα έβλεπες, γιατί δεν βλέπεις τη διαφορά. Και αυτό είναι το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που άρχισα λίγο να καταφτάσω στην αίθουσα. Ε, δεν ε, άκουσα δηλαδή ε, την παρουσίαση δυστυχώς, αλλά άκουσα τη συζήτηση που έγινε. Και δεν θέλω τώρα να ε, ε, έτσι να είμαι δικηγόρος του διαβόλου, δεν θέλω από την άλλη πλευρά να αρχίσουμε να συζητούμε τους ε, δείκτες τους οποίους θέλουμε να συμπεριλάβουμε μέσα στο κανονισμό. Αλλά από την άλλη πλευρά δηλαδή θα πρέπει να πω ότι το γεγονός ότι έχουμε τόσους πολλούς δείκτες μέσα στον, ε, στους κανονισμούς ε, που ισχύουν σήμερα αποτελεί μια μεγάλη τροχοπέδηση ό,τι αφορά την ε, αξιοποίηση αυτών των κοντιλίων. ακριβώς δηλαδή αυτή η υψηλή γραφειοκρατία είναι που εμποδίζει τελικά την απορρόφηση των κοντιλίων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε σε περιφερειακό επίπεδο. και η Μόνικα να το ανέφερε δηλαδή ότι έχουμε καταφέρει να επιβάλλουμε τη διάσταση του φύλου ω οριζόντιο κριτήριο και μέσα στον κανονισμό των γενικών διατάξεων. Όταν λοιπόν εμεί συζητούμε εδώ, εντάξει, καλώ ε, τα συζητούμε, ε, και δεν ξέρω και κατά πόσο αν θα είχαμε καταφέρει να λάβουμε υπόψη και τι προτάσει που κάναμε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν δεν είχαμε επιμείνει σε ό,τι αφορά ακριβώ το οριζόντιο κριτήριο μέσα στο κείμενο του κανονισμού. Αλλά από την άλλη πλευρά, υπενθυμίσουμε εδώ ότι εμεί στο Κοινοβούλιο είχαμε ταχθεί υπέρ ε, αυτού του στοιχείου. Δηλαδή, α μην νομίζει κανεί ότι τα κράτη-μέλη είναι πολύ υπέρ όλων αυτών των προοδευτικών ιδιών που εμεί ε, προτείνουμε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το βλέπω δηλαδή και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν ε, χώρα τώρα με τα κράτη-μέλη. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να επιτύχουμε κάποια πρόοδο σε ό,τι αφορά ε, τα ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το Κοινοβούλιο, όπω αυτό εδώ το ζήτημα τη διάσταση τη ισότητα των φύλων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε τα πορίσματα από αυτή τη μελέτη να μεταφερθούν και στι διάφορε περιπέτειε, να μην παραμένουν μόνο εντό στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου ακριβώ να υπάρξει περισσότερη ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Δεν ωφελεί δηλαδή σε τίποτα να συμφωνούμε εμεί σε επίπεδο θεσμικών οργανώτου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να αναλυφθεί η δράση. Όχι, στι ίδιε τι περιοχέ, εκεί λαμβάνει η χώρα τελικά η υλοποίηση των προγραμμάτων. Και δεν μπορούν και οι διαχειριστικέ αρχέ, τα managing authorities να επιτύχουν τα πάντα. Όχι, θα πρέπει δηλαδή όλοι όσοι εργάζονται εκεί σε αυτό το περιφερειακό επίπεδο και όσοι έχουν και οικονομική αρμοδιότητα να το λαμβάνουν αυτό υπόψη τους ε, ε, και στο πλαίσιο του ΙΤΕΣ για παράδειγμα και στο ε, Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξη, για παράδειγμα, χρειαστήκαμε χρόνια έτσι ώστε σιγά σιγά πράγματι να εδραιωθεί αυτή η διάσταση και η λήψη υπόψη τη διάσταση των φίλων Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορούμε εμεί απλώ να αποφασίσουμε και να διατάζουμε από την πλευρά των Βρυξελών. Θα πρέπει αυτή η προσπάθεια να μεταφερθεί στι ίδιε τι ε, περιφέρειε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε για παράδειγμα με την Επιτροπή των Περιφερειών και με έπαφε με τι ίδιε τι περιφέρειε. Ε, για παράδειγμα με, ε, με, με επικοινωνία και, και με γραπτή επικοινωνία, για παράδειγμα, με τα διάφορα περιφερειακά ε, κοινοβούλια, τι διάφορε επιτροπέ σε περιφερειακό επίπεδο, ε, προκειμένου ακριβώ να ληφθούν υπόψη τα πορίσματα αυτή τη μελέτη. Δηλαδή, αυτό, αυτή η προσπάθεια, αυτή η προσέγγιση θα μα ωφελήσει. Δεν θα μα ωφελήσει απλώ και μόνο η προσθήκη περαιτέρων δικτών μέσα στον ε, κανονισμό. Και κάτι τέτοιο άλλωστε δεν θα μα ωφελούσε γιατί ήδη έχουμε παγιώσει την ε, θέση μα ως κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά ε, το νέο κανονισμό. Νομίζω πως εκείνο που θα πρέπει λοιπόν να γίνει και εκείνο που έχει πιο πολύ νόημα είναι να υπάρξει περισσότερη ευαισθητοποίηση στο επίπεδο των περιφερειών προκειμένου η ίδια η νοοτροπία αν θέλετε στι περιφερειε να λαμβάνει πλέον υπόψη τη διάσταση του φίλου. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Κωνσταντς, που μας τιμήσατε αυτή την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποφύγει τις ευθύνες που έχει επί του ζητήματος αυτού. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων ε, έδωσε το Κοινοβούλιο μάχη για, τις, για την εξάντερη σημότητα όπως και για τις αρχές ε, των εταιρικών σχέσεων. Σήμερα εξακολουθούμε να δίνουμε μάχη, να αγωνιζόμαστε για τον σεβασμό των αρχών αυτών, αλλά είναι αλήθεια και η μελέτη σας το δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των ε, χωρών και μεταξύ των περιφερειών ως προς την πραγματικότητα αυτή. Περιμένουμε από την Επίτροπο όταν αναλάβει τα καθήκοντά της να υλοποιήσει τις αξίες και τις αρχές αυτές και ίσως αυτό αναφέρθηκε και σε μία από τις παρεμβάσεις και νομίζω ότι η Μελλοντική Επιτροπή θα είναι και αρμόδια για θέματα μεταρρύθμισης και ελπίζω να έχει μία προοδευτική στάση στην προσέγγιση αυτή και όχι να μιλούμε απλώς για την υλοποίηση διαρθωτικών οικονομικών μέτρων και ίσως στη μεταρρύθμιση και με την υποστήριξη που μπορεί να δώσει η Επιτροπή στα κρατημέλη, θα χρειαστεί να ενσωματωθούν και αυτές οι διαστάσεις του σεβασμού των αρχών αυτών. Μας αναφέρατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με τις πολύ σημαντικές στην πραγματικότητα δυνατότητες που έχουμε για την υποστήριξη της ισότητας των δικαιούχων των μέσων συνοχής στα πλαίσια του Ταμείου Ανάπτυξης Υπέθρου. Τα ακούσαμε όλα αυτά, τα σημειώνουμε, έχουμε μεγάλη δουλειά, μεγάλη προσπάθεια ακόμα να κάνουμε, αλλά έχω και ένα ερώτημα που είναι ίσως, ε, ακούγεται ίσως ως λίγο παράδοξο. Αναφέρεστε σε μια ανησυχία σχετικά με πιθανές οπισθοδρομίες στο μέλλον, σχετικά με την ισότητα των φύλων στα κράτη και τις περιφέρειες. Ωστόσο έχουμε την εντύπωση καμιά φορά ότι το θέμα αυτό σήμερα είναι ένα θέμα που διαρκώς δηλώνουν ως ε, πολιτική προτεραιότητα οι διάφοροι ηθήνοντες. Το ακούμε στις, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια στις συζητήσεις μας και εδώ και 10 ε, χρόνια θα έλεγα δεν συζητούμε πλέον δεν το εξετάζουμε δηλαδή. Είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα ω προτεραιότητα ισότητα των φύλων σε όλε τι χώρε και λέω τι περιφέρειε. Και επομένω υπάρχουν σίγουρα δυσκολίε στην εφαρμογή, στην υλοποίηση. Και αυτό είναι το στοιχείο που θα πρέπει να παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ εκ νέου για τη μελέτη σα. Ευχαριστώ του συναδέλφου για την πλούσια ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Και θα παρακαλούσα να πάμε τώρα στο, σημείο, στο επόμενο σημείο της διατάξεως. Ευχαριστώ. Nous passons à présent. Ας πάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως. στα πλαίσια του οποίου θα ήθελα να, καλωσορίσω την κυρία Μαρία Νακότσεβα. Je Σας ευχαριστώ κυρία Γενική Διευθυντή της Eurostat για την παρουσία σας εδώ σήμερα το απόγευμα. Εδώ και κάποιες εβδομάδες είχαμε την ετήσια έκθεση για τα στατιστικά, στατιστικά δεδομένα των περιφερειών διανεμήθηκε από την Eurostat. Εμείς το παρακολουθούσαμε με μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να μπορέσει να σας ακούσει σήμερα. Σας καλωσορίζω και πάλι και σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Η στατιστική ενημέρωση τα στατιστικά δεδομένα είναι θεμελιώδες εργαλείο ώστε να αξιολογούμε τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων ε, στο έδαφος, των προγραμμάτων των έργων. Και εσείς ασχολείστε με τη συλλογή στατιστικών δεδομένων πανευρωπαϊκών, εθνικών αλλά και περιφερειακών τοπικών. Για την περιφερειακή διάσταση, οι στατιστικές αυτές αναλύσεις πραγματοποιούνται από τα κράτη-μέλη από τα κράτη-μέλη υπό το ΝΑΤΣ, την αρχή των, των τριών αυτών επιπέδων στατιστικών ε, στοιχείων, δεδομένων. Η Eurostat έχει διευκρινίσει, έχει συγκεκριμενοποιήσει τα στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιεί, ώστε να μην βασίζεται μόνο στον αριθμό των κατοίκων, αλλά σε συγκεκριμένες περιφέρειες, σχετικά με αστικές μονάδες, παράκτιες, νησιωτικές, ορεινές κτλ. Διαφορετικά λοιπόν στοιχεία που είναι πολύτιμα για εμάς και που μας δίνουν μια συνολική πληροφορία για την ε, κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή την οποία έχει ως αντικείμενο να υλοποιεί και επανεξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε τρία χρόνια. Κυρία Κότσεβα, λοιπόν, σας προσκαλέσαμε εδώ για να μας παρουσιάσετε τη δουλειά της δικής σας υπηρεσίας και του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να συνεισφέρετε στην επεξεργασία των πολιτικών μας. Αλλά και επίσης για να μας περιστέσετε συνολικά την ετήσια έκθεση 2019. Ε, διάβασα με μεγάλη προσοχή εγώ το έγγραφο και όπως κάθε χρόνο νομίζω ότι μπορούμε σταδιακά να έχουμε μια όλο και πιο εξειδικευμένη απεικόνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύτιμων στατιστικών στοιχείων για την κοινωνική πρόνοια, για τις διαφορές της ψηφιακής τεχνολογίας που διατίθεται στους πολίτες των διαφόρων χωρών. Μία δηλαδή χαρτογράφηση των κενών που υπάρχουν στις περιφέρειες στην εδαφική μας συνοχή. Και που η Ευρωπαϊκή μας Επιτροπή έχει ως αντικείμενο ως στόχο να, τα, να τις καλύψει, να καλύψει αυτά τα κενά, αυτές τις ελλείψεις. Θα ακούσουμε λοιπόν την παρουσίασή μας και μετά θα ακούσουμε τα μέλη για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Εμείς χρησιμοποιούμε κυρίως τα αγγλικά στο Eurostat. Ετοιμάζουμε συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για όλο τον κόσμο επίσης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά για μένα αυτή και τιμή μου που έχω τη δυνατότητα να σας μιλήσω. Τα στατιστικά στοιχεία κατά την άποψή μου είναι σωστή χρήση. Αν δεν χρησιμοποιούνται τα στατιστικά στοιχεία είναι ατελής η αποστολή μας. Γι' αυτό είναι σημαντικότατο να γίνονται αυτού του είδους παρουσιάσεις. Το είπατε άλλωστε. Να δείξουμε τι κάνουμε. Να πάρουμε το έντυπο το πρόσφατο με τα περιφερειακά στοιχεία, να παρουσιάσουμε και τι άλλε υπηρεσίε που παρέχουμε όσον αφορά τα στοιχεία και να ανταλλάξουμε απόψει μαζί σα, κυρίω σχετικά με το πώ θα θέλετε να χρησιμοποιήσετε τι πληροφορίε, πώ τι βρίσκετε τι πληροφορίε, τι είναι σημαντικό. Απόλαυσα την προηγούμενη παρουσίαση. Ήρθα εκεί που στο τέλο συζητούσατε τη σωστή προσέγγιση για την ε, προσμέτρηση των ανισοτήτων, πώς η διάσταση του φύλου μπορεί να ενταχθεί στα στατιστικά στοιχεία. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Αισθανόμουν πολύ οικία όταν άκουγα την προηγούμενη συζήτηση. Ξεκινώ με την παρουσίαση. Ετοιμάστηκε από την ομάδα της Eurostat. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι εντό της παρουσίασης. Είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε μετά να διερευνήσετε το θέμα περαιτέρω και αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Να πω καταρχάς ότι όλα τα στοιχεία βλέπετε το λογότυπο του στατιστικού του Eurostat που είναι η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είναι σημαντικό για τη Eurostat που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχουμε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι είμαστε τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τη DG Regio με την οποία συνεργάζεται στενά. Το άλλο σκέλος της Eurostat είναι στα κράτη-μέλη, διότι το Eurostat δεν παράγει τα στοιχεία μόνο του. Το Eurostat συνεργάζεται με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Αυτό είναι κατανοητό. θέλουμε ερωτηματολόγια να κάνουμε έρευνες και αυτά πρέπει να γίνονται στο τοπικό επίπεδο και γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά με εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Και αυτό που σας παρουσιάζω είναι ένα κοινό προϊόν της στατιστικής κοινότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Eurostat αποτελείται από 800 μέλη και οι στατιστικολόγοι στα κράτη-μέλη είναι 50.000. Ακόμα και αυτά τα στατιστικά στοιχεία για μας σας δείχνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα εσάς γιατί τα στατιστικά στοιχεία που παράγουμε είναι σημαντικότατα. Εδώ με σύγχρονο τρόπο, με εικόνες παρουσιάζουμε διάφορα παραδείγματα χρήσης στατιστικών στοιχείων, πολιτική συνοχής, Φερρυπίν, ξεκινώντας από εκεί. Όταν θέλω εξηγήσω στα παιδιά μου τι κάνω όταν δεν είμαι στο σπίτι που λείπω συνέχεια να καταλαβαίνουν πιο εύκολα. Τους λέω ότι βάσει των στοιχείων της Eurostat και κυρίως βάσει περιφερειακού ΑΕΠ κατά κεφαλή, κατά άτομο, σε συγκρίσιμη αγοραστική ισοτιμία, αυτό δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λέω τώρα βέβαια, αλλά αντιλαμβάνονται τέλο πάντων τα στοιχεία όσον αφορά το ΑΕΠ χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ή την περιγραφή των λιγότερων επιτυγμένων περιφερειών εκεί που το ΑΕΠ τους είναι λιγότερο από 75% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η αφετηρία για την περίοδο 2014 2022, όταν ξεκινήσαμε. Να δούμε ποιες είναι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές για να δούμε σε ποιο πληθυσμό στοχεύουμε. Και βάσει άλλων δικτών εφαρμόζονται άλλες πολιτικές. Για το Ταμείο Συνοχής, το, ακαθο... το καθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ένα άλλο στατιστικό στοιχείο οικονομικής α, επίδοσης. Και υπάρχουν και άλλες συγκεκριμένες πολιτικές που γίνονται σημαντικότερες και γι' αυτό αλλάζουν οι απαιτήσει για στοιχεία. Πρόσφατα, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση, η ανάπτυξη της υπαίθρου και σχετική πολιτική, το θεματολόγιο της πόλης, Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, αποτελούν αναδιόμενες ε, ανάγκες για στοιχεία. Και τώρα στο παγκόσμιο προσκήνιο, το θεματολόγιο του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα άλλο ευρύ πλαίσιο όπου η Eurostat παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο παράγοντας εκθέσεις εποπτικές όπου εκεί βλέπουμε πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους στόχους του 2030. Και υπάρχει ένας στόχος, ο στόχος 11 νομίζω, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν ε, την περιφερειακή ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάσατε άριστα ένα τμήμα των διαφανειών μου όταν είπατε ότι όλα τα περιφερικά στατιστικά στοιχεία βασίζονται στον ορισμό. Τι εννοούμε όταν λέμε περιφέρεια περιοχή. Και έχουμε το ακρονίμιο NUTS που προέρχεται από τα γαλλικά καθορίζει ε, περιφερειακές μονάδες, εδαφικές μονάδες και αυτή είναι η βάση. Χρόνια συζητούν οι στατιστικολόγοι κάποιους ορισμούς θα σας δώσω παράδειγμα σε επόμενες διαφάνειες τι δεν έχουμε επιλύσει ακόμα ως ορισμό. Και στον κόσμο καν. Εδώ έχουμε τις περιφερειακές μονάδες. Κάθε χώρα υποδιαιρείται σε τρία επίπεδα περιφερειών. Ένα, δύο και τρία. Ένα είναι μεγαλύτερη μονάδα, δύο η επόμενη και τρίτη είναι η μικρότερη. Βασίζονται επί πληθυσμιακών κριτηρίων, όπως αναφέρατε, το 1, η περιφέρεια Notch 1 είναι ανάμεσα στα 3 και 7 εκατομμύρια κατοίκους, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιες χώρες όπως είναι η Εστονία, η Λετωνία, η Μάλτα, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο έχουν μόνο μια περιφέρεια. Νοτ 1. Σε όρους Ευρωπαϊκής Ενώσεως ΝΑΤΣ 2 είναι οι περιοχές από 800.000 μέχρι 3 εκατομμύρια κατοίκους και ΝΑΤΣ 3 είναι ανάμεσα στις 150.000 και 800.000 ανθρώπους. Ε, δεν χρειάζεται να, να θυμόσαστε του αριθμούς, θα πρέπει να θυμόσαστε ποια είναι η βάση αυτών των περιφερειών που για τις πολιτικές βασίζεται η κατάταξη σε αριθμό κατοίκων. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Τι πρέπει να ξέρετε για την ταξινόμηση όταν αναλύετε τα στοιχεία. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές οι περιοχές, αυτές οι περιφέρειες αντιστοιχούν επίσης σε διοικητικές περιφέρειες, αφετηρία είναι το ΝΑΤΣ 3, το χαμηλότερο επίπεδο, και μετά κινούμεθα στο ανώτερο επίπεδο, ομαδοποιώντα, προσθέτουμε διοικητικέ περιοχέ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι χρησιμοποιούνται και άλλα κριτήρια πέραν των αριθμητικών. Ε, βάζουμε και διοικητικό κριτήριο που αφορά την εφαρμογή της πολιτικής. Κάτι άλλο σημαντικό. Έχουμε λάβει σχετικά ερωτήσεις, όπως και εσείς πάνω σε αυτό πόσο άκαμπτη είναι η ταξινόμηση, πόσο θα μπορούσαμε να αλλάξουμε ταξινόμηση. Αναφέρεται στον κανονισμό ότι δεν μεταβάλλονται πιο συχνά από κάθε τρία χρόνια. Παραμένει η ταξινόμηση για τρία χρόνια και κάθε τρία χρόνια ζητάμε από τα κράτη-μέλη να μας πούν κατά πόσο έχουν διαπιστώσει κάποιες αλλαγές λόγω αλλαγής του πληθυσμού ή λόγω διοικητικών μεταρρυθμίσεων και μετά πρέπει να μας ενημερώσουν. Ελέγχουμε κατά πόσο τα κριτήρια, η λογική πίσω από όλα αυτά πίσω την ταξινόμηση είναι η σωστή και μετά συνδυάζουμε όλες τις εκθέσεις των κρατών μελών και έτσι έχουμε τη νέα επικαιροποιημένη εκδοχή που παρουσιάζεται. Η παρούσα εκδοχή είναι του 2016. Τι σημαίνει αυτό? Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι καθορίζουμε τον κατάλογο των περιφερειών στο τέλος του 2016. Τέλος, είναι στο τέλος του εγχειριδίου και όταν καθορίσουμε τις περιφέρειες, τότε τα, ε, τα κράτη έχουν ένα χρόνο να προσαρμοστούν αν κάτι πρέπει να γίνει και αρχίζουν μετά τον επόμενο χρόνο να υποβάλουν πληροφορίες. Οπότε το το 2016, η ταξινόμηση αυτή το 2016 περιέχει στοιχεία που ξεκίνησαν να υποβάλλονται το 2018 και το βιβλίο αυτό, το εγχειρίδιο που βλέπετε, που δημοσιεύτηκε, αντικατοπτρίζει στα στοιχεία που παραθέτει τη νέα ταξινόμηση. Μην, μην περιμένετε επαναστάσεις. Ε, υπάρχει σχετι... μεγάλη σταθερότητα, ελάχιστες αλλαγές ε, με την πάροδο των ετών στις περιφέρειες. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα διαφάνεια. Η προηγούμενη διαφάνεια αναφερόταν στις περιφέρειες που είναι κοντά στη διοικητική δομή των χωρών, αλλά αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή και όπως είπατε, και λόγω των αναγκών της πραγματικής ζωής και λόγω πολιτικών προτεραιοτήτων υπάρχουν διαφορετικές περιφερειακές διαστάσεις που ταιριάζουν με δικαιτικές. Οι πόλεις, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε πόλεις. Έχουμε το αστικό θεματολόγιο. Τι χρειάζεται λοιπόν απόλυτα. Να έχουμε περιφερειακά στοιχεία για τις πόλεις, να καθορίσουμε τι εστί πόλεις ποιοι μετακινούνται προς και από την πόλη. Και γι' αυτό θα πρέπει να καθορίσουμε και το κέντρο της πόλης, αλλά και τους ανθρώπους που πηγαίνουν έρχονται για να εργαστούν στην πόλη, που αποκαλείται αυτό λειτουργική αστική περιοχή. Στατιστική ορολογία χρησιμοποιώ, που δεν μπορεί να σας λέει τίποτα, αλλά γι' αυτό είναι σημαντικό α, να έχουμε απλές εξηγήσεις. Όταν προσθέτεις στην πόλη τους εργαζόμενους απ' έξω από την πόλη έχει τη λειτουργική αστική περιοχή. Όταν προσθέτεις και στο κέντρο της πόλης τις περιφερειακές διοικητικές μονάδες, έχεις ευρύτερη πόλη ή μητροπολιτική περιοχή. Ένα παράδειγμα. Μιλάνο. Ρίχνα μια ματιά τώρα, τον ερχόμενο το Λουξεμβούργο. Το Μιλάνο έχει περίπου 1.300.000 ε, κατοίκους. Αν προσθέσεις κανείς και αυτούς που έρχονται για να εργαστούν στο Μιλάνο, φτάνει στα 5 εκατομμύρια κατοίκους. Τρεις φορές παραπάνω δηλαδή. Αν δεν θέλεις να λαμβάνεις υπόψη μόνο αυτούς που εργάζονται αλλά τη διοικητή περιοχή γύρω από τους Δήμους, από το Μιλάνο, που είναι από όπου έρχονται οι περισσότερο 50% από τους μετακινούμενους, φτάνει στο 4 εκατομμύρια, στο νούμερο αυτό θα πρέπει να έχουμε στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο πόλης, μητροπολιτικής περιοχής, σε επίπεδο μετακινούμενων εργαζομένων, διότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές που εξαρτώνται από αυτό, υποδομές μεταφορικές, δημόσιες μεταφορές κλπ. Αυτού του είδους στατιστικά στοιχεία που βασίζονται επί τέτοιου είδους τυπολογίες, όλο και περισσότερο ε, σημαντικά γίνονται. Παρομοίως είχαμε και ορισμό των περιοχών της υπαίθρου, της υπαίθρου βασίζεται στην πυκνότητα του πληθυσμού ορισμός αυτός και επί της ε, του πληθυσμού κλπ. Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις της ζωής και αν έχουμε κάποιο έργο τα επόμενα χρόνια να κάνουμε είναι να συμπληρώσουμε τα παραδοσιακά στατιστικά στοιχεία των τυπικών περιοχών ΝΑΤΣ, των κλασικών περιοχών ΝΑΤΣ, με στατιστικά στοιχεία που παράγονται βάσει των νέων ε, τυπολογιών, δεσυνοριακές περιοχές, παράκτης περιοχές, πόλεις υπαίθριες περιοχές όπου χρειάζεται στοιχεία για να μπορείς να εφαρμόζεις τις πολιτικές. Αυτό είναι το ιστορικό. Πάμε στα προϊόντα. Είναι σαν ένα μενού για σας. Να σας δείξουμε τι μπορούμε να σας δώσουμε στα στοιχεία και ελπίζουμε ότι στην ανταλλαγή απόψεων, μέσω ανταλλαγής απόψεων θα μπορέσετε να δείτε τι μπορούμε να σας δώσουμε. Λοιπόν, έχουμε αυτό, αυτή τη βίβλο μας ούτως είπε, είναι ένα χειρίδιο Έχουμε τρεις βίβλους, τρία τέτοια έντυπα, ετήσια τεστικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εγχειρίδιο. Δεύτερο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο σε σύγκριση με τις άλλες χώρες και ένα εγχειρίδιο ε, περιφερειακά στοιχεία της Eurostat. Δεν ξέρω αν με πιστεύετε, αλλά είναι και το πιο σημαντικό αυτό και το πιο ζητούμενο διότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία. Ενδιαφέρεται ο κόσμο για τι περιφέρειε, είναι πιο κοντά στου πολίτε τη περιφέρεια, είναι σημαντική περιφέρεια τη πολιτική. Άλλη περιφερειακή διάσταση υπάρχει σε διάφορα στατιστικά στοιχεία, αλλά είναι πολύ δύσκολο να πάει κανεί σε διάφορε περιοχέ. Είναι πιο δύσκολο δηλαδή κάποιο να αναζητά τι επιμέρου ε, περιφερειακέ ε, συλλογέ ε, από το να έχει συγκεντρωμένα τα στοιχεία στην στο, στο, στο ίδιο υλικό και να μπορεί δηλαδή να κάνει τις διάφορες συνδέσεις ε, που χρειάζεται. Ε, μπορεί λοιπόν ε, κανείς ε, να ε, κατεβάσει την όλη επιτηρίδα, το όλο εγχειρίδιο ή μπορεί να το κάνει ένα κεφάλαιο. Εδώ βλέπετε την διάθρωση των διαφόρων κεφαλαίων. Έχετε λοιπόν τα περιφερειακά δεδομένα για όλες αυτές τις περιοχές που βλέπετε. Μιλάμε δηλαδή για παιδεία γενικά, με μεγάλο εύρος και εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι το βασικό επίπεδο στο οποίο δημοσιεύονται τα σχετικά στατιστικά δεδομένα είναι το επίπεδο NATS 2, δηλαδή στατιστική εδαφική μονάδα 2. Γιατί αυτό είναι το αρχικό επίπεδο σύλλογης αυτών των δεδομένων. Και από εκεί και μετά, πέραν αυτής της δομής ε, που έχουμε μέσα σε αυτήν την επιτρέπεια, έχουμε και δύο διαφορετικά, κάθε χρόνο διαφορετικά, ε, σημεία η παιδεία ε, στα οποία δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση. Για την φετινή, για παράδειγμα, έκδοση έχουμε από τη μία την εστίαση στις ευρωπαϊκές πόλεις και από την άλλη την εστίαση ε, στις ε, περιφερειακές κοινωνικονομικές εξελίξεις. Βέβαια, ο τίτλος είναι πολύ γενικόλογος, ε, και το αντιλαμβάνομαι, αλλά από την άλλη πλευρά για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά ακριβώ αυτέ τι εξελίξει στι κοινωνικονομικέ περιφέρειε, ο στόχο είναι να βλέπουμε ακριβώ το ποιε είναι οι εξελίξει που λαμβάνουν ε, χώρα σε βάθο χρόνου. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τι αγροτικέ περιοχέ. Τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη δημογραφική σύνθεση των ανθρώπων που διαμένουν στι αγροτικέ περιοχέ. Λοιπόν, οι περιφέρειε λοιπόν διέρχονται ορισμένε αλλαγέ. Λαμβάνουν χώρα, υπάρχουν κάποιε τάσει οι οποίε παρατηρούνται. Οπότε, με τέτοιου είδου εστίαση που κάνουμε, δίνουμε κάποια ρεθίσματα για σκέψη ω προ το τι συμβαίνει και πώ μπορεί με αυτόν τον τρόπο να μετεξελιχθεί η χάραξη πολιτική. Εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα μας, ε, όταν για παράδειγμα έχετε μπροστά σα, είτε στην έντυπη μορφή του, είτε σε μορφή PDF ε, το εγχειρίδιο την ευετρίδα μας. ε, βλέπετε εδώ κάποιου χάρτες οι οποίοι είναι πολύ ενδεικτικοί και σας δίνω τρία ε, παραδείγματα σε αυτές τις τρεις διαφάνειες. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι οι χάρτε είναι πολύ σημαντικοί σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά στατιστικά δεδομένα, γιατί ακριβώ περνούν το μήνυμα με πολύ απλό τρόπο. Η συγκεκριμένη διαφάνεια έχει να κάνει με τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Και πάλι μιλάμε για επίπεδο ΝΑΤΣ 2. Και βλέπετε σε διαφορετικά τώρα χρώματα του τι συμβαίνει στι διάφορε περιφερειε. Όπω θα θυμόσαστε, ένα από του στόχου τη στρατηγική 2020 ήταν να μειωθεί ο αριθμό αυτών των ατόμων, δηλαδή εκείνων που εγκαταλείπουν πρόωρα ε, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και να φτάσουμε σε επίπεδο κάτω από το 10%. Μιλάμε δηλαδή για άτομα τα οποία καταλήγουν προώρα ειδικότερα το σχολείο. Βλέπουμε λοιπόν σε μπλε χρώμα τις περιοχές οι οποίες έχουν επιτύχει αυτόν τον στόχο, δηλαδή του λιγότερο από 10% του συνόλου για τα άτομα εκείνα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ενώ σε ε, πορτοκαλί για παράδειγμα βλέπουμε ε, τις περιοχές εκείνες και χωρίς όπου δεν έχουμε επιτύχει το απαραίτητο επίπεδο και απέχουμε. Βλέπουμε λοιπόν πολύ εύκολα ε, με μια ε, ματιά στο χάρτη το πού θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες. Επίσης εκείνο που είναι σημαντικό είναι το ότι βλέπουμε διαφορετικές διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές περιοχές μέσα στην ίδια χώρα. Άρα λοιπόν για την ίδια χώρα υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές σε ό,τι αφορά τι επιμέρου ε, περιφέρειε. Για παράδειγμα, στην Ουγγαρία βλέπουμε να υπάρχουν ακριβώ τόσο μεγάλε διαφοροποιήσει. Δηλαδή, βλέπουμε όλε τι διάφορε χρωματικέ αποχρώσει στην ίδια χώρα. Το ίδιο ισχύει για τη Βουλγαρία. Όπου δηλαδή ε, ε μόνο μία περιοχή επιτυχεί τον ε, απαραίτητο στόχο, ενώ όλε οι άλλε περιοχέ υστερούν. Τώρα, επόμενη διαφάνεια, άλλο παράδειγμα, πάλι με χάρτη, σε ό,τι αφορά το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανακάτοικο. Βλέπετε λοιπόν σε όλη την Ευρώπη ποιες είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες έχουν, βρίσκονται πιο κοντά στον, ε, στον μέσο όρο, ποιες είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένε για παράδειγμα σε μπλε χρόνο και εκείνες που ε, υστερούν περισσότερο. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η τάση ε, σε ορισμένες ε, χώρες... Ε, υπάρχει εστίαση της οικονομικής ανάπτυξης, ε, για παράδειγμα, στη ε, Μπρατισλάβα ή, στην, για παράδειγμα, στην Πολωνία, στη Βαρσοβία και ούτω καθεξής. Δηλαδή, εστίαση της οικονομικής ανάπτυξης στις περιοχές των πρωτεύουσων. Πολύ δηλαδή κεντρική ανάπτυξη, όπου έχουμε έναν υδροκεφαλισμό τη πρωτεύουσα, όπου λαμβάνει η χώρα όλη η οικονομική ανάπτυξη εκεί. Και από εκεί και μετά έχουμε άλλε χώρε όπου ακριβώ λαμβάνει η χώρα η οικονομική ανάπτυξη σε διαφορετικά κέντρα. Και δεν έχουμε ιδιαίτερη εστίαση δηλαδή εκεί σε μια περιοχή. Αυτό για παράδειγμα παρατηρείται και στη Γερμανία και στην Ιταλία. Αυτό βέβαια για να επιτευχθεί προϋποθέτει και διαφορετικές οικονομικές πολιτικές. Ένα ακόμα παράδειγμα που θα σας δώσω σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που έχουμε σε χάρτες είναι το επίπεδο απασχόλησης αναπεριοχή. Και πάλι βλέπουμε εδώ εύκολα στο χάρτη ποιε είναι οι περιοχέ, ποια είναι τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν επιτύχει τους στόχου του 2020, δηλαδή 75% ποσοστό απασχόλησης. Και εδώ είχα κρατήσει τη σημείωση για μένα ότι αυτό που θα πρέπει να πω και στην ομάδα μου ότι θα πρέπει να έχουμε και εδώ διαφοροποίηση και διαχωρισμό φύλου. Δηλαδή θα πρέπει να βλέπουμε εδώ το επίπεδο απασχόλησης είτε, ε, είτε για τους άντρες είτε για τις γυναίκες. Ε, ήταν ε, πολύ σημαντική λοιπόν η προηγούμενη παρουσίαση που έγινε ακριβώ σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Αυτό σε ό,τι αφορά λοιπόν την επιτελεία, το yearbook και το τι περιλαμβάνει αυτό. Και Ε, αυτή τη διαφάνεια θα την προσπεράσω και θα σας την ε, παρουσιάσω τελευταία. Να σας εξηγήσω λοιπόν ποια είναι τα άλλα εργαλεία επικοινωνίας που έχουμε με το κοινό. Πέραν από το yearbook, την επετρίδα, υπάρχουν και περαιτέρω εργαλεία ε, που είναι πολύ χρήσιμα για την εργασία σας και ε, για να τα βρείτε μπορείτε να μπείτε μέσα από την πύλη μας το Eurostat ε, και ελπίζω να λειτουργεί βέβαια κανονικά η πύλη εδώ, δεν τη δοκίμασα τώρα τελευταία αλλά σίγουρα θα τη βρείτε. Εδώ λοιπόν αν κάνετε μια αναζήτηση θα φτάσετε στην αρχική σελίδα της Eurostat και εκεί λοιπόν για τις ε, ειδικότερες περιοχές και τις ε, πόλεις μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα διαφορετικά εργαλεία σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που σας συναφέρω και θα εστιάσω σε κάποια από αυτά που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Το πλέον χρήσιμο εργαλείο που θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε στην καθημερινή σας εργασία είναι το εργαλείο My Region, η περιοχή μου, η περιφέρεια μου. Καταρχήν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο iPhone σας ή και στον υπολογιστή και μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα τη δική σας περιφέρεια. Και, δηλαδή την εκλογική σας περιφέρεια. Να ε, επιλέξετε λοιπόν τους δείκτες που σας ενδιαφέρουν για τη δική σας περιφέρεια και αυτομάτως λαμβάνετε μια παρουσίαση αλλά και μια σύγκριση της περιφέρειάς σας με τον υπόλοιπο κόσμο. Και πράγματι ε, εδώ έχουμε συμπεριλάβει τους δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνότερα, δηλαδή που έχουμε λάβει σχολιασμά από εσά ότι του αξιοποιείτε και του έχετε ανάγκη περισσότερο. Αλλά βέβαια είμαστε ανοιχτοί και σε προτάσει, γι' αυτό χρειαζόμαστε και feedback και σχόλια. Ο στόχο μα βέβαια δεν είναι να σα ε, πλημμυρίσουμε με χιλιάδες διαφορετικούς δείκτες, θέλουμε να σας παρέχουμε τους δείκτες εκείνους, τους οποίους έχετε ιδιαίτερη ανάγκη και τους χρησιμοποιείτε επανειλημμένα όταν μεταβαίνετε στις εκλογικές σας περιφέρειες, όταν επικοινωνείτε με, τους, ε, με το εκλογικό σα. σώμα. Δηλαδή, να μπορείτε εύκολα να ανοίγετε το iPhone σας ή να ανοίγετε την εφαρμογή, να επιλέγετε την περιφέρειά σας και να λαμβάνετε άμεσα τα πιο σημαντικά σταχεία που σας ε, ενδιαφέρουν. Τώρα, ένα διαφορετικό εργαλείο με διαφορετικό είδος παρουσίας είναι το Regions and Cities Illustrated, δηλαδή απεικόνιση των περιφερειών και των πόλεων. Ε, στο προηγούμενο εργαλείο είχαμε λοιπόν στοιχεία για τη δικιά σας ε, την περιφέρεια και σύγκριση αυτών των στοιχείων με τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ έχετε το σύνολο ε, της Ένωσης ή ε, της Ευρώπης και επιλέγετε το συγκεκριμένο θέμα το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο για το οποίο λαμβάνετε πληροφορίες σε ό,τι αφορά όλες τις ε, περιφέρειες. Βλέπετε λοιπόν εδώ το χάρτη, το γράφημα και τα διάφορα στοιχεία τα οποία βέβαια δεν είναι αναγνωστά εδώ στη διαφάνεια. Με βάση λοιπόν μπορείτε με αυτά τα στοιχεία να κάνετε δική σας ανάλυση, ή να κατεβάσετε το χάρτη, να κατεβάσετε τα στοιχεία και ούτω καθεξής, αλλά αυτά είναι πιο τεχνικά ζητήματα και αφορούν κυρίως τους ε, εμπειρογνώμονές σας, τους βοηθούς σας ε, και ούτω καθεξής. Ε, πάντως πρόκειται για στοιχεία δηλαδή τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν για να κάνετε περαιτέρω ανάλυση. Ε, στο κάτω εδώ μέρος πάντως μπορείτε να δείτε ένα χρονοδιάγραμμα εδώ με διαφορετικά έτη. Κάνοντας λοιπόν κλικ σε κάθε έτος μπορείτε να δείτε την δυναμική εξέλιξη σε βάθος χρόνου και βλέπετε πώς εξελίσσεται δηλαδή ο χάρτης σε βάθος χρόνου. Και αυτό πάλι μπορεί να σας ε, δώσει περισσότερα ρεθίσματα για το πώ μπορείτε να διεξάγετε περαιτέρω αναλύσει. Ένα τρίτο εργαλείο ή τρίτο προϊόν είναι ο στατιστικό χάρτη, Statistical Atlas, που τα λέει όλα δηλαδή, είναι ένα στατιστικό χάρτη ακριβώ. Ε, σε αυτό εξυπηρετεί και περιλαμβάνει ουσιαστικά όλους τους χάρτες τους οποίους σας δείξαμε ήδη και στο πλαίσιο της παρουσίας της επαιτρίδας. Ε, μεταβαίνετε λοιπόν ευθεία με την επιλογή που κάνετε στο χάρτη σε ό,τι αφορά με συγκεκριμένη ε, περιφέρεια ή μια συγκεκριμένη περιοχή ή ένα συγκεκριμένο θεματικό πεδίο και μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το χάρτη έτσι ώστε να ενσωματώσετε αυτό το υλικό στην, ε, στη δουλειά σας. Τώρα, τι έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε κατά τελευταία 2-3 χρόνια προσπαθούμε να διευκολύνουμε τη δουλειά των χρηστών μας. Ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παραπονεθεί επανειλημμένα και συμφωνώ με αυτό το παράπονο ότι ε, η, η πύλη μας είναι πολύ χρήσιμη για τους ερευνητές ε, αλλά όχι για τους ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερη γνώση των ζητημάτων και θέλουν να βρουν τα δεδομένα ε, που του ενδιαφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν, ε, ε, ακριβώ για να διευκολύνουμε αυτή τη δουλειά, για εκείνου που δεν έχουν αυτέ τι τεχνικέ γνώσει, έχουμε συμπεριλάβει κάποια βίντεο tutorials, δηλαδή κάποια βίντεο ε, που δίνουν οδηγίε ω προ το τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε λοιπόν και μέσα σε λίγα λεπτά σα δίνετε ακριβώ καθοδήγηση ω προ το τι μπορείτε να βρείτε πού σε ό,τι αφορά στατιστικά δεδομένα της Eurostat. Και από εκεί και μετά υπάρχουν και πιο παραδοσιακοί, αν θέλετε, τρόποι ενημέρωση. Δηλαδή, με βάση τις ε, μελέτες που έχουν γίνει, ένα απλό ενημερωτικό δελτίο, το newsletter δηλαδή, και απλά δεδομένα ε, που διανέμονται ε, στους χρήστες, πραγματικά μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά εργαλεία. Και πριν από δύο εβδομάδε λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή την έκδοση ενημερωτικού δελτίου, newsletter. Είναι πολύ πρόσφατο, μόνο λοιπόν μία έκδοση έχει εκδοθεί και μέσω αυτή προσπαθούμε να ενημερώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα του χρήστε μα ποια είναι τα πιο πρόσφατα εργαλεία μας, ποιε είναι οι πρόσφατες εξελίξεις, ποια είναι η ενημέρωση των ε, στατιστικών στοιχείων που έχουν γίνει, ε, ποιοι χάρτες και κάνουμε και κάποιους διαγωνισμούς δηλαδή σε ό,τι αφορά το, τα δεδομένα του μήνα, το χάρτη του μήνα ε, και από εκεί και μετά μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε μέσω ακριβώ τη σελίδα τη Eurostat για να λαμβάνετε το newsletter. Επίση είμαστε πολύ ενεργοί στα μέσα κοινωνική, δικτύωση στα social media Facebook και Twitter γιατί θεωρούμε πως αυτά είναι τα μέσα τα οποία ενδιαφέρουν τους νέους οι οποίοι ακριβώς θέλουν να λαμβάνουν απλά στατιστικά στοιχεία και αυτό το αντιληφθήκαμε κι εμείς. και γι' αυτό, επειδή συνήθω είναι σε αγγλική γλώσσα τα γραφήματα τα οποία δημοσιεύουμε, είναι πάντοτε απλά έτσι ώστε να είναι και απλή η μετάφρασή του στι διάφορε ε, ε, γλώσσε. Ε, και υπάρχουν δηλαδή ε, φορείς ε, στα διάφορα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται πολύ να λαμβάνουν αυτά τα απλά γραφήματα έτσι ώστε απλά να μπορούν να τα μεταφράζουν και στην εκάστοτε γλώσσα. Και αυτό είναι και ένα από τους τρόπους ε, που μπορούμε να επιτύχουμε ακριβώς περισσότερη εγκύτητα με το κοινό μα. δηλαδή μετάφραση αυτών των στοιχείων στι εκάστοτε γλώσσες έτσι ώστε μπορούμε να έχουμε καλύτερη επαφή με τα κοινά ανά με το κοινό ανά μέλος. Αν θέλετε τώρα περισσότερη υποστήριξη, έχουμε και θεσμική υποστήριξη, institutional support από πλευρά τη Eurostat. Υπάρχει εδώ μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, ε, μέσω τη οποία μπορείτε να έρθετε προσωπικά σε μαζί μα, αλλά υπάρχει και γραφείο μα εδώ στι Βρυξέλλε, γιατί βέβαια τα κεντρικά μα γραφεία τη Eurostat βρίσκονται στο Λουξεμβούργο. Ε, βρισκόμαστε λοιπόν στη διάθεσή σα, ε, έτσι ώστε να σα παράσουμε ad hoc δυνατότητες δηλαδή να λάβετε δεδομένα που σας ενδιαφέρουν. Στο τέλος εδώ της παρουσίασης σας έχω συμπεριλάβει links ε, συνέσμους δηλαδή με όλα τα στοιχεία τα οποία σας ε, παρουσίασα μόλις τώρα. Και επανέρχομαι τώρα στην ε, παρουσίαση την οποία δεν αποφάσισα να σας παρουσιάσω τελευταία, δηλαδή ως προς το τι ακριβώς θα κάνουμε μελλοντικά. Μελλοντικά λοιπόν τα περιφερειακά δεδομένα θα καταστούν όλο ένα και πιο σημαντικά. Ποια είναι λοιπόν η βασική πρόκληση εδώ ε, για μας και ποια υποστήριξη θέλουμε να λάβουμε από τη δική σας πλευρά. Όταν κανείς θέλει να εμβαθύνει περισσότερο την ανάλυση του στις επιμέρους δηλαδή μικρές περιοχές και θέλουμε ταυτόχρονα να υπάρχει ε, η ανάλυση σε ό,τι αφορά δηλαδή τη δημοκρατική σύνθεση, φύλλο και ούτω καθεξής Από τη μία πλευρά λοιπόν χρειάζονται και περισσότερες ε, έρευνες ευρύτερε, με περισσότερε δαπάνε και ούτω καθεξή. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και οι νέε τεχνολογίε οι οποίε μα επιτρέπουν και εναλλακτικού τρόπου συγκέντρωση των δεδομένων. Υπάρχει το επωνομαζόμενο geocoding. Και έχουμε για παράδειγμα τι γεωεδαφικέ συντεταγμένες για παράδειγμα και για τις πόλεις και ε, τις ε, περιοχές. Και προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε ε, για κάθε κτίριο τις γεωσυντεταγμένε και σε ό,τι αφορά του ανθρώπου που διαβιώνουν και, και αυτό γιατί. Γιατί μόλι κανεί έχει τις συντεταγμένε, μπορεί να ορίσει κανεί ω περιοχή που τον ενδιαφέρει οτιδήποτε. Μπορεί για παράδειγμα να είναι ένα πολεοδομικό τετράγωνο, μπορεί να είναι μια ευρύτερη περιοχή, μια τονιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για παράδειγμα σε ό,τι αφορά εμ, παρεμβάσει, σε ό,τι αφορά αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών εμ, ε, και ένα σώρο άλλε σοβαρέ πολιτικέ. Και αυτή είναι η μεγάλη μα φιλοδοξία μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Να είμαστε σε θέση δηλαδή να παρέχουμε πιο λεπτομερή περιφερειακά στοιχεία χρησιμοποιώντα ακριβώ γεωεδαφικά δεδομένα σε συνδυασμό με στατιστικά δεδομένα. Και από εκεί και μετά υπάρχει μια απογραφή ε, πληθυσμιακή δηλαδή που θα λάβει η χώρα πανευρωπαϊκά το 2021 και είναι είναι η μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο στατιστικό εγχείρημα το οποίο θα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής ε, και μέσω του οποίου ελπίζουμε να έχουμε περισσότερα δεδομένα αξιοποιώντας ακριβώς και αυτόν τον συνδυασμό στατιστικών και γεωγραφικών δεδομένων. Ε, συνεργαζόμαστε λοιπόν στενά και με την DG Regio και τι υπόλοιπε υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το επιτύχουμε, αλλά χρειαζόμαστε τη συνεργασία ε, και τη δική σα ήδη. Συνεργαζόμαστε καλά, χρειαζόμαστε και την υποστήριξη των υπηρεσιών γεωχαρτογράφησης, geomapping. Και εκεί ακριβώς θέλουμε και περισσότερη συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές αρχές και θέλουμε να ακουστούν και οι δικές σας φωνές, δηλαδή από την πλευρά των χρηστών μας, ότι πραγματικά έχετε ανάγκη ε, αυτά τα δεδομένα. Γιατί μόνο εφόσον υπάρχει αυτή η ανάγκη και είναι ξεκάθαρη. Μπορούμε και εμεί να δικαιολογήσουμε το γιατί κάνουμε αυτά που κάνουμε, γιατί εμβαθύνουμε περισσότερο τα περιφερειακά δεδομένα. Αυτά από την πλευρά μου και βέβαια θέλω να ακούσω τι δικέ σα απόψει γιατί πρόκειται για ε, μια δυναμική ε, εξέλιξη εδώ όπου συνέχεια αναπροσαρμόζουμε τα όσα προσφέρουμε λαμβάνοντας υπόψη τα όσα χρειάζεται εσείς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τι δικέ σα απόψει. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Merci. Ευχαριστούμε την κυρία Κότσεβα για την ε, παιδαγωγικότατη αυτή η παρουσίαση που μας έκανε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Πεκάρινεν. Ευχαριστώ κυρία Γενική Διευθυντά. Με ενθαρρύνεται, λέει ο μιλητής, να χρησιμοποιήσω την μητρική μου. Θα μιλήσω λοιπόν στα φιλανδικά. Ήθελα λοιπόν καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. γιατί μας κάνατε μια πληρέστατη εισαγωγή ε, για το σύστημα στατιστικών δεδομένων των ε, περιφερειών και τι ακριβώς παρέχει. Θα ήθελα να καταλάβω λίγο πιο συγκεκριμένα εκεί όπου έχετε κάποιες εσαλληλουχίες χρονικές για τους δείκτες εκείνους οι οποίοι ε, δείχνουν ποια, ποιο είναι το καθεστώς της περιφερειακής ανάπτυξης. Στη δημοσίευσή σας υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά δεδομένα, τα οποία καταδεικνύουν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εσείς λοιπόν χρησιμοποιείτε αλληλουχίες χρονικές οι οποίες δείχνουν την επιτυχία της προσπάθειας ή την πρόοδο των ε, πολιτικών συνοχής Έχετε λοιπόν χρονικές αλληλουχίες για το ΝΑΤΣ 3. Και γιατί ε, χρειαζόμαστε αυτές τις ε, χρονικές αλληλουχίες για το ΝΑΤΣ 3 για την κοινή ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών μονάδων 3 βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περιπτώσεις ε, ολόκληρης χώρας που βρίσκεται στην αυτή περιοχή ΝΑΤΣ. Βλέποντας όμως τα, δεδομένα του ΑΕΠ και ονομαστικά, αλλά και σε σχέση με τον μέσο όρο της ε, ε, ανάπτυξης της υπαίθρου στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι οι περιοχές ΝΑΤΣ 3 εκτός των μεγαλοναστικών κέντρων έχουν μείνει σταθερές ή και έχουν ελαφρά μειωθεί σε κάποιες περιπτώσεις και σε σύγκριση με τον ενωσιακό μέσο όρο. Εσείς λοιπόν παράγετε αυτές τις χρονικές αλληλουχίες που θα μας επέτρεπαν να έχουμε μία πιο λεπτομερή χαρτογράφηση, απεικόνηση του πώς δαπανώνται τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για να γνωρίζουμε και πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η πόρη σε επίπεδο περιφερειών. We are discussing how I should <laughs> now. Ε, συζητούσαμε με τον Πρόεδρο πώς θα έπρεπε να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ καλή σας ερώτηση. Υπάρχουν δύο στοιχεία που θα ήθελα να σχολιάσω. Καταρχάς αυτές οι χρονικές αλληλουχίες. Το μειονέκτημα της ε, έντυπης δημοσίευσης είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε τρισδιάστατες, τρισδιάστατα γραφήματα και επίσης πρέπει να καλύπτουμε και όλες τις περιφέρειες. Ε, εξού και τα ψηφιακά μέσα είναι τα καλύτερα γιατί μπορεί να είναι διαδραστικά και να μπαίνει σε χρονικέ αλληλουχίε. βεβαίω και τι χρησιμοποιούμε. Το θέμα είναι σε ποιο επίπεδο και για ποιου δείκτε. Τα πιο χρησιμοποιημένα επίπεδα, ιδιαίτερα στου οικονομικού δείκτε στου οποίου αναφέρεστε, είναι στο ΝΑΤΣ 2. Στο επίπεδο ΝΑΤΣ 3 είναι, αν θέλετε, ο επόμενος στόχος, θα μπορούσα να πω. Γιατί δεν έχουμε όλους τους δείκτες στο επίπεδο ΝΑΤΣ 3. χρονικές αλληλουχίες σίγουρα έχουμε στον ΝΑΤΣ 2 και αν δείτε και την τράπεζα δεδομένων της ε, Eurostat είναι προσβάσιμα αυτά τα δεδομένα. Τώρα αναφερθήκατε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή σχετικά με την χρονική εξέλιξη ή πρόοδο της εφαρμογής των πολιτικών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναφέρθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση. τι δείκτες θα μπορούσαμε να, παράγα, να παράγουμε ώστε να εξασφαλίζουν μια καλύτερη παρακολούθηση της προόδου των πολιτικών. Είναι μια συζήτηση που διεξάγεται και με το ελεγκτικό συνέδριο, για παράδειγμα, σχετικά με το πώς ποσοτικά απεικονίζουμε τις επιδόσεις. Εμείς συλλέγουμε τις πληροφορίες, αλλά πρέπει να γίνει μια συζήτηση, μια πλήρη συζήτηση με εμπειρογνώμονες αξιολόγησης πολιτικών συνοχής. Εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια τέτοια συζήτηση, αλλά ως στατιστικοί οι δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, αν θέλετε, επί του συσχετισμού συγκεκριμένων παρεμβάσεων και των αλληλουχιών που βλέπετε. Εμείς πάντοτε συνιστούμε να είστε προδραστικοί, να συζητήσετε συζητάτε με τους ηθήνοντες πολιτικής, να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που επιθυμείτε να καταμετρήσετε, προκειμένου εμείς να σας προτείνουμε τους καλύτερους δείκτες για αυτό. Επομένως και η Eurostat παίζει, διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση ή στην ανάπτυξη τέτοιων δικτών στους οποίους αναφέρεστε και ήταν πολύ καλό χρονικό σημείο εκείνο της ερώτησής σας πριν από το επόμενο ΔΕΛΤΑΠΗ γιατί θα πρέπει να ρυθμίσουμε και όλη τη δομή μας, τους μηχανισμούς μας για να συλλέξουμε τα απαραίτητα εδωμένα και υπό απαραίτητο ή κατάλληλο μορφότυπο. Ναι, λέει ο Πρόεδρος, κοιτάξτε. Το ελεκτικό συνόδριο το οποίο θα ακούσουμε αύριο ε, έθεσε ακριβώς το ερώτημα κριτηρίων αξιολόγησης των επιδόσεων της περιφερειακής πολιτικής. Είναι πραγματικά ένα, θέμα, ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Ο κύριος Πάντζα έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλό απόγευμα σε όλες ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κυρία Κότσεβα για την πολύ καλή παρουσίαση. Είναι ένα εργαλείο που είναι εξαιρετικά πολύτιμο, χρήσιμο για εμάς, τα μέλη του Κοινοβουλίου, στο Μιλάνο, πόλη στην οποία ζω, αποτυπώνονται η διάδραση που υπάρχει μεταξύ του αστικού κέντρου, του Μητροπολιτικού κέντρου και της υπόλοιπης ε, περιφέρειας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Στην εδαφική κατανομή ή στην εδαφική αξιολόγηση που γίνεται μεταξύ αστικών κέντρων και παρακτήων περιοχών, για παράδειγμα. Υπάρχει ένας σχετισμός ε, στον οποίο προβαίνει και το Κοινοβουλίο και η Κομισιόν, αλλά λείπει ε, ε, το στοιχείο, της, το στοιχείο του κατακόρυφου, οι ορεινές περιοχές. Ίσως ζητώ συγγνώμη δηλαδή από τους συνοδέλφους που έχουν ήδη συζητήσει το θέμα αυτό, αλλά επειδή εγώ προέρχομαι από ορεινή περιοχή, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Γιατί δηλαδή δεν λαμβάνουμε υπόψη το στοιχείο του κατακόρυφου. Έχουμε τρεις περιφέρειες ε, στην Ιταλία, Μπελούνα, Σόντριο και άλλη μία, που το Ιταλικό κράτος θεωρεί περιφέρειες ιδιαίτερα ορεινού χαρακτήρα, οι οποίε δεν μπορούν να συγκρίνονται με άλλες περιφέρειες υπαίθρου, λόγω της γεωγραφίας τους ή δεν μπορούν να συγκριθούν με παιδινές περιοχές στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Μιλούμε για τελείως διαφορετικά προβλήματα, τελείως διαφορετικό ανάγλυφο απαιτήσει και ιδιαιτερότητες. Και καθότι μιλούμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο και για μια πιο προσεκτική ε, μέθοδο γεωεντοπισμού των δεδομένων, δεν θα έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη μας και αυτήν την ιδιαιτερότητα γιατί η Ιταλία πράγματι έχει όλο το αλπικό ανάγλυφο αλλά και άλλες χώρες η Αυστρία είναι απολύτως ορεινή χώρα η Ελβετία είναι εξ ολοκλήρου ορεινή οι Γαλλικές Άλπεις ε, τα Πυρηναία πολλές περιοχές ε, στην Ευρώπη που είναι αντίστοιχες, αντίστοιχης ιδιαιτερότητας. Ήθελα να καταλάβω λοιπόν αν στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα λαμβάνουμε υπόψη μας, θα προσέχουμε λίγο κάποιες περιοχές που είναι ναι της υπαίθρου αλλά είναι πολύ διαφορετικές από άλλες παιδινές. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Χαίρομαι που τυχαία πέλεξα το παράδειγμα του Μιλάνου. Δεν είμαι ειδικό για να μπορέσω να αξιολογήσω την ε, φύση της πολιτικής που εφαρμόζεται. Κατά πόσο αυτές οι περιοχές, οι ορεινές περιοχές, θα πρέπει ε, να είναι ειδικό αντικείμενο πολιτικής παρέμβασης και πώς συσχετίζονται με την ύπεθρον γέννη. Να σας απαντήσω από πλευρά στατιστικής. Είναι ένα έξοχο παράδειγμα αυτό που παραθέσατε, που επιβεβαιώνει γιατί θα πρέπει να έχουμε ε, γεωεντοπιστικά στοιχεία, στοιχεία που ιστορικά εξατώνταν από τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων. Και η συλλογή των στοιχείων εξαρτάται από διοικητικές δομές, σε κάποιο βαθμό. Όταν δημιουργήσαμε τις περιφέρειες και καταρτήσαμε την κατανομή ΝΑΤΣ, ξεκινούσαμε πάντα από διοικητικές οντότητες που θα μπορούσαν να συλλέξουν τα στοιχεία. Δήμους, μεγαλύτερες περιοχές, κράτος, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα ακολουθούσαμε τη διοικητική δομή, δεν είχαμε άλλη δυνατότητα συλλογή στοιχείων. Αλλά αν έχουμε γεωχωρικά στοιχεία, ε, τότε εμείς σαν στατιστικολόγοι μπορούμε να έχουμε μια βάση που είναι σημαντική. Και αν είχατε γεωλογική κωδικοποίηση, μπορούσατε να ομοδοποιήσετε στοιχεία και να θέσετε όπως επιθυμείτε τεχνικώς πώς τα όρια. Αυτός είναι ο στόχος. Να μπορούμε να έχουμε τέτοιο πλούτο στοιχείων και ευελιξία, να έχετε τις κατάλληλες πληροφορίες, την κατάλληλη βάση για να πάρετε μετά αποφάσεις για την κατάλληλη πολιτική, βάση κοινωνικών ε, παραγόντων, πολιτικών παραγόντων, τι είδους απόφαση πρέπει να λάβετε. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό όταν έχετε την απογραφή του πληθυσμού και ξέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά των πολιτών, εάν υπάρχει και γεωλογική κωδικοποίηση των στοιχείων, μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε υποδιέρεση θέλετε. Γι' αυτό η τεχνική μας φιλοδοξία είναι να μπορούμε να παρέχουμε τις βασικές πληροφορίες που θα σας επιτρέπουν να ε, αποφασίζετε κατάλληλα μετά από την κατάλληλη συζήτηση για την εφαρμοστέα πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αντρέι Νοβάκοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Κότσεβα, σας συγχαίρω για την παρουσίασή σας και για τη δουλειά που έχετε κάνει. Εντυπωσιάστηκα. Λέγοντας το αυτό, ομολογώ ότι ομιλίες για τα στατιστικά στοιχεία στο Πανεπιστήμιο ήταν από τα αγαπημένα μου θέματα. Ε, δημιουργήσατε κατατίσατε, ετοιμάσατε ένα πολύ καλό έγγραφο. Έχω μια πλούστατη λύση για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Μπορούμε να έχουμε ε, επίσης και το yearbook, αυτό υπό οποιαδήποτε μορφή. Χάρτινη έκδοση, ηλεκτρονική, απλούστατο. Ναι, φέραμε κάποια αντίγραφα της επετηρίδας αυτής. Αν θέλετε, μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερα αντίγραφα ψηφιακά. Μπορούμε να σας δώσουμε το σύνδεσμο να κατεβάσετε το έγγραφο. Ζούμε σε καιρούς όπου οι πληροφορίες είναι πολυτιμότατες. Εποχές όπου οι ψευδείς δύσεις ε, είναι πληθώρα. Χρειαζόμαστε επιστημονική βάση, στοιχεία που μπορούμε να εμπιστευτούμε για τις αποφάσεις μας. Αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε στο Facebook και στο Twitter παρουσιάζοντας στοιχεία απλά, εικόνες απλές, στατιστικές που να μπορεί και ο απλός άνθρωπος να καταλάβει. Πολύ καλή ιδέα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω αυτό. Συνεχίστε, συνεχίστε, καλά πάτε. Η σχέση μας, ενώ εσείς από πλευρά Eurostat και εμείς από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα στη σχέση αυτή. Θα πρέπει τακτικά να μας ενημερώνετε για να είμαστε ενήμεροι για το μέλλον. Είσαστε ένας από τους μεγαλύτερους στατιστικούς φορείς στον κόσμο. Πρέπει να αποφεληθούμε από αυτό. Κυρίως στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καθημερινά εργαζόμαστε με βάση αυτά. Περιφέρειες, οικογένειες, πόλεις, χώρες, επίπεδο Νότστρια, Επιχειρήσει, σχολεία, πολιτική συνοχής, καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωή του ανθρώπου. Πρέπει να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας. Με διευθυντές σαν και εσάς μπορούμε να τα καταφέρουμε, να τα πάμε πολύ καλά και να κινηθούμε και πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Αντρέι Νοβάκοφ. Πράγματι δίκιο έχεις. Γι' αυτό θέλαμε το απόγευμα να διεξαχθεί αυτή η ακρόαση. Αληθεύει επίσης ότι θα πρέπει στο μέγιστο βαθμό να αναπτύξουμε τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων και της Eurostat. Λοιπόν, τα στατιστικά ε, στοιχεία αφορούν πολύ την πολιτική μας την περιφερειακή. Και οι ελάχιστες πολιτικές είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένες με τα στατιστικά στοιχεία, διότι οι δικές μας πολιτικές εδράζονται επί κατηγοριών περιφερειών που συνδέονται αυτές με τη σειρά τους με τα στατιστικά στοιχεία και τα στοιχεία που παράγεται και η αλλαγή αυτών μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες ως αφορά τις αποφάσεις μας για διάφορα θέματα που άπτονται το επικέντρο της περιφερειακής πολιτικής. Τα στοιχεία που παράγεται λοιπόν έχουν αντίκτυπο συγκεκριμένο και αποτελέσματα. Και γι' αυτό προφανώς η Eurostat είναι ένας εταίρος σημαντικότατος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Επιτροπή μας, τη Ρέτζη, όλος ιδιαίτερος και είσαστε ο φορέας εκείνος που από τους ε, πρώτους ε, έρχεται εδώ για να συμβάλλει στην ακρόαση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νοβακόφ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, εξαιρετική σας πανεβασία γιατί η δική μου παρουσίαση εστιάστηκε σε αυτά που χρειάζεστε εσείς. Αλλά ο, ρόλος που μπορεί να παίξει η Eurostat από κοινού με άλλα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των fake news είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα προσωπικά και εδώ βασίζομαι ε, στο, στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε συνέργειες μεταξύ μας, χρειαζόμαστε συνεργασίες ε, και θα πρέπει ε, να έχουμε για τα δεδομένα μας, για παράδειγμα, fact-checkers, δηλαδή εκείνους από την πλευρά των μέσων ενημέρωσης, από την πλευρά του Κοινοβουλίου, θα ελέγχουν ακριβώς τι ειδήσει ω προ το αν είναι αληθή, βασιζόμενοι και στα ε, δεδομένα που εμεί παρέχουμε. Και αυτό, για παράδειγμα, στο πλαίσιο, για παράδειγμα, τη προεκλογική εκστρατεία για τι ευρωεκλογέ, δημιουργήσαμε ακριβώ μια τέτοια συνεργασία με διάφορου fact-checkers, ακριβώ, παρέχοντα ιδιαίτερη υπηρεσία, μέσω της οποίας μπορούσαν να λαμβάνουν 24 ώρες υποστήριξη από τη δική μας πλευρά για να τους απαντούμε ερωτήματα σε ό,τι αφορά δεδομένα προκειμένου να διευκολυνθεί όλη η συζήτηση που γινόταν προεκλογικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σα σχόλιο, ε, πριν από κάποιους μήνες δημιουργήσαμε μια συνεργασία με, το, με την ερευνητική σας υπηρεσία του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την παροχή συγκεκριμένων ε, δεδομένων και θεωρώ πως ε, εδώ θα πρέπει να διευθύνουμε αυτή τη συνεργασία μας και με το Γραφείο Επικοινωνίας του Κοινοβουλίου γιατί δεν υπάρχει τίποτα ισχυρότερο από το να περιλαμβάνετε τα, την, Eurostat, τα στοιχεία μας στις δικές σας δημοσιεύσεις, στα δικά σας ε, tweet. Ε, ειδικότερα αξιοποιώντα τη δυνατότητα μετάφραση ε, των δεδομένων μα σε όλε τι γλώσσε τη Ένωση. Είμαστε λοιπόν πεπισμένοι ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτονόητο το ότι οι άνθρωποι θα μεταφέρουν στην ιστοσελίδα τη Eurostat για να βρουν τα δεδομένα που του ενδιαφέρουν. Θα πρέπει να του βοηθήσουμε και θα σας πω κάτι το οποίο είναι το δικό μου όνειρο και ίσως να σας ακουστεί αστείο, αλλά επειδή εγώ ταξιδεύω πολύ, γιατί έχω πολλές ε, ε, διεθνείς συναντήσεις για να έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα και ούτω καθεξής, ε, συχνά έχω συνομιλίες ε, με οδηγούς σε ταξί και εκείνοι με ρωτούν τι δουλειά κάνω και τους λέω εργάζομαι για γύρω Eurostat και τι μου λένε, τι μου απαντούν Ε, συνέχεια μπερδεύουν ε, την Eurostat με την Eurostar και, μας λένε, και μου λένε οι οδηγοί ταξί, μα τα τρένα σας είναι συνέχεια αργοπορημένα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το όνειρό μου. Όταν μία μέρα θα μπαίνω σε ένα ταξί και θα με ρωτάει ο οδηγό τι δουλειά κάνω και θα του λέω ότι δουλεύω για την Eurostat, θα την αγνωρίζει και θα μου λέει Α, ναι, ε, χθε είδα κάποιο, κάποιο δεδομένο, κάποιο στοιχείο που με ενδιέφερε ε, και θα αναφέρεται στην Eurostat και δεν θα την μπερδεύει με την Eurostat και δεν θα μου λέει ότι τα τρένα σα αργούν συνέχεια. Θα ήθελα λοιπόν μία μέρα η Eurostat να αποτελέσει το σημείο αναφορά για τα στατιστικά δεδομένα σε όλη την Ευρώπη. Ελπίζω να έρθει αυτή η μέρα ε, και χαίρομαι πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να ε, συνομιλούμε, να συζητούμε για το πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ μα Γιατί έχουμε μια κοινή αποστολή εδώ, την οποία υποστηρίζουμε και το Κοινοβούλιο και η Eurostat. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ απολύτως βεβαίως σχετικά με τη σημασία των δεδομένων που μας παρέχεται. και θα είχε υπάρξει αδύνατον για εμάς να υπερασπιστούμε την σημασία της πολιτικής συνοχής όταν είχε αμφισβητηθεί χωρίς να έχουμε αυτά τα δεδομένα. Εγώ, Γενική Διευθυντή, ε, προέρχομαι από τη Ρουμανία και στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε ένα πολύ πολύ σημαντικό ε, μεταναστευτικό πρόβλημα. <coughs> Περισσότερα παιδιά ε, των πολιτών μας γεννιόνται εκτός της χώρας παρά εντός της χώρας. Έχουμε ένα μαζικό μεταναστευτικό ρεύμα προς τα έξω. Εδώ μπορεί να συζητήσει κανείς την ε, σημασία ή την αποτελεσματικότητα των μέσων της πολιτικής συνοχής, ε, το πόσο πρέπει να τα υποστηρίξουμε και άλλο ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά αλλά κυρίως πρέπει να εστιαστούμε και στο πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τους πολίτες της περιφερειάς από τις οποίες προέρχονται. Και, πολύ σημαντικό εδώ είναι το θέμα των θέσεων απασχόλησης, αλλά πάνω απ' όλα των θέσεων απασχόλησης με αξιοπρεπή μισθό. Διότι διαφορετικά φεύγουν οι πολίτες. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στη Ρουμανία, συνολικά στην Ανατολική Ευρώπη λέει ο μιλητής. Δηλαδή άνθρωποι με πανεπιστημιακό επίπεδο μόρφωσης αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες και προβλήματα στη χώρα τους και επομένως λαμβάνουν την απόφαση να φύγουν και αφήνουν πίσω τους ένα κενό. Στη Ρουμανία έχουμε πάρα πολλά έργα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε διότι έχουμε χάσει τους άνθρωπινους πόρους που μας χρειάζονται προκειμένου να τα υλοποιήσουμε. Αυτή λοιπόν, αυτό το φαινόμενο της μετανάστευσης πλήττει ιδιαίτερα τις ε, ε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και έχω και μια ε, γνωμοδότηση ιδίας πρωτοβουλία ε, και στην Άγκρη αλλά και στην Ρέγκη συζητείται ιδιαίτερα αυτό. Δεν ξέρω λοιπόν αν εσεί είχατε κοιτάξει αυτό το ιδιαίτερο θέμα. Ε, και φαίνεται να υπάρχει μια απόκληση ως προς τα φύλλα σε αυτό το επίπεδο. Ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο είναι η μετανάστευση των γυναικών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης γιατί σε σχέση με αυτό το ε, φαινόμενο μετανάστευση πολλά παιδιά, μικρά παιδιά αφήνονται πίσω, χωρίς τη φροντίδα τη μητέρα τους και αντιμετωπίζοντα πολύ μεγάλη δυσκολία ώστε να ενταχθούν τελικά μεγαλώνοντα στο παραγωγικό ιστό της χώρας. Εμεί έχουμε και νέα κυβέρνηση στη Ρουμανία, πάρα, πάρα πολύ πρόσφατα, και θα μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να καταλάβουμε πώ αποτελεσματικά θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά να εφαρμόσουμε πολιτικέ που θα μπορέσουν να κρατήσουν του πολίτε μα εντό τη χώρα και να συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο στην συνολική ανάπτυξη ή πρόοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει η προοδο Σα ευχαριστω πολυ Κότσεβα και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό από την εμπειρία μου σε εθνικό επίπεδο στατιστικής και τώρα πλέον σε ευρωπαϊκό και έχω και ούτως ή άλλως και ένα ακαδημαϊκό παρελθόν σε αυτό το πεδίο, το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι πραγματικά, ε, αν θέλετε, είναι ένα πρόβλημα του πώς μπορεί κανείς να αντλήσει στατιστικά δεδομένα, ήδη σχετικά με το πρόβλημα αυτό εθνικά, πολύ περισσότερο δεν περιφερειακά. Εκεί λοιπόν έχουμε μια σημαντική πρόκληση του πώς ποσοτικά θα καλύψουμε αυτό το μέγεθος, ιδιαίτερα στον παραδοσιακό τρόπο ανάπτυξης ή παραγωγής στατιστικών δεδομένων που είναι πανεθνικά. Χρειάζεται όμως να έχουμε μια ανταλλαγή πληροφοριών, ενημέρωσης, δεδομένων με τις χώρες που περισσότερο αφορά το, φαινόμενο αυτό, όπως η δική σας η χώρα, η Βουλγαρία, χώρες που αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικό φαινόμενο διασποράς προς το Ηνωμένο Βασίλειο, προς την Ισπανία ή την Ιταλία. Χρειάζεται λοιπόν μια ανταλλαγή στατιστικών δεδομένων μεταξύ των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών της χώρας προορισμού και προέλευσης. Και είναι δύσκολο διότι υπάρχουν και διάφορες διατάξεις ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων μεταξύ άλλων αλλά μερικές φορές ακόμα και ανταλλάσσοντας μεγέθη απλώς αριθμών, αναφύλλο, αναμορφωτικό επίπεδο κτλ. μας βοηθούν να έχουμε μια ακριβέστερη εικόνα του μεταναστευτικού φαινόμενου, αλλά οφείλουμε ακόμα προς την κοινωνία να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα σε αυτό το φαινόμενο. Συμφωνώ μαζί σας. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και θα επισκεφθώ και τον Ιανουάριο το Βουκουρέστι διότι η κυβέρνησή σας θέλει να εξετάσει τις ε, νέες τεχνολογίες σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου μετανάστευσης. Θα, το, θα συνεργαστούμε και με την Παγκοσμία Τράπεζα, ιδιαίτερα για χώρες όπως της Ανατολικής Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο έντονης φυγής. Και ελπίζω να μπορέσουμε να προοδεύσουμε, αλλά πράγματι δεν είναι εύκολο εφόσον δεν ανταλλάσσετε εσείς δεδομένα με τις χώρες προς τις οποίες μεταναστεύουν οι πολίτες. Στο κανονισμό έχετε συζητήσει πολλούς, στο κοινοβούλιο με συγχωρείτε, έχετε συζητήσει πολλές διατάξεις κανονισμών ανταλλαγής δεδομένων, αλλά πολύ συχνά έχουμε προβλήματα με την ιδιωτικότητα των δεδομένων, αλλά έχουμε τη σταθερή δυσκολία ανταλλαγής μεταξύ χωρών για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την απάντηση, ακριβέστατη απάντηση. Κίκας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Έχω ερώτηση. Όχι την ομαδοποίηση των στοιχείων, αλλά τη χρήση. Τη μετέπειτα. Είπε σωστά και ο Σαντρα Νοβακόφ ότι είσαστε ένας από τους μεγαλύτερους φορείς συλλογή στοιχείων, παραγωγής στοιχείων. Έχω την εντύπωση ότι χρησιμοποιείτε ο φορέας σας λάθος. Σαν να έχεις πολύ καλό υπολογιστή και χρησιμοποιείς τον υπολογιστή σας σφυρί για να καρφώνεις καρφί στον τοίχο. Ο υπολογισμός του ΑΕΠ είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Πρωτόγωνο θα έλεγα, αρχικό στοιχείο. Εσείς σαν στατιστικολόγος ίσως να μην είσαστε ικανοποιημένοι που έχετε σαν βασικό στοιχείο το ΑΕΠ. Λαμβάνονται υπόψη πολλοί αόριστοι παράγοντες. Δεν είναι πολύ καλή εκτίμηση. Η Eurostat έχει εναλλακτική όσον αφορά το ΑΕΠ να δείχνει βαθμό, βαθμό ευημερίας, αύξηση της ευημερίας και άλλες ε, πτυχές. Από ΑΕΠ θα κινηθείτε προς άλλο παράγοντα, άλλο δίκτυο. Ή θα κρατήσετε το ΑΕΠ μέχρι ότου ληφθεί μια διαφορετική πολιτική απόφαση. Και αν ισχύει αυτό, θα υποστηρίζατε την αλλαγή από ΑΕΠ προς κάποιον άλλο δίκτυ. Έχετε κάποιες ιδέες. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η αλλαγή, τι θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, εμπεριείχε πολλές στοιχές. Έχουμε πολλά στοιχεία στη διάθεσή μας στο Eurostat. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Βασική μου συμβουλή είναι ότι αν θες μια πλήρη εικόνα, πώς να το πω, η τέχνη έγκυται στο να βρεις την πληροφορία που θα σου αποκαλύψει την όλη εικόνα. Σχετικά με αυτό, θέλαμε να ενισχύσουμε τη χρήση των στοιχείων Eurostat για έρευνα σε επίπεδο πολύ μικρό, πολύ λεπτόμερες ή να δώσουμε δυναμικά εργαλεία που μπορούν να συνδυαστούν και να μπορεί ο χρήστης να αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αντικειμενικά. Όσον αφορά το ΑΕΠ, ακόμα και τώρα δεν είναι ο μόνος δείκτης επί του οποίου με βάση φάση του οποίου λαμβάνονται υποφάσεις για την πολιτική συνοχή. Υπάρχουν μετά και θέματα εφαρμογής προγραμμάτων και υπάρχουν διάφοροι δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται. Κοινωνικοί δείκτες, απασχόληση, ανεργία φερρυπίν, επίπεδο παιδείας, δεν χρησιμοποιείται μόνο το ΑΕΠ. Αυτή είναι η απάντησή μου θα έλεγα. Και τώρα η μορφή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, η διαμόρφωσή της εδώ θα πρέπει να λαμβάνει χώρα. Μαζί με το Συμβούλιο και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτούς τους διαλόγους η Eurostat γιατί, γιατί μπορούμε να σας πούμε τι είναι προσμετρήσιμο και τι δεν είναι. Κάποιοι θέλουν να υπολογίσουν το ΑΕΠ Φερρυπίν του οδούς στην οποία μένω. Ε, δεν αστειευόμαι. Αυτή είναι ακραία περίπτωση. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει κάποιος δίπλα σου που να σου περιγράφει τι είναι εφικτό, τι είναι προσμετρήσιμο, τι δεν είναι. Καμιά φορά ο δείκτης μπορεί να είναι ένα πολύ καλό θεωρητικό οικοδόμημα, αλλά στην πράξη να μην μπορεί να συλλέξει τα στοιχεία. Διότι αυτό είναι το ζουμί. Να συλλέξει τα στοιχεία στην πράξη. Αν στείλει ένα ερωτηματολόγιο με 100.000 ερωτήσει, κανεί δεν θα απαντήσει το ερωτηματολόγιο και θα πάει στη σωστή απάντηση. Άρα δεν έχει σωστή εικόνα. Αυτέ είναι ακραίε περιπτώσει. Αλλά έχουμε πληροφορίε, έχουμε δείκτε. Πώ τα χρησιμοποιούμε το θέμα. Και πώς μπορούμε να προσμετρήσουμε τη σωστή διανομή των πόρων, αυτό είναι κάτι προ συζήτηση των εμπειρογνωμόνων. Δεν είναι ένα καθαρό στατιστικό θέμα και στατιστικό καθήκον. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρέμβαση. Ο κύριος Τέλειος Κιμπουρόπουλος. Ε, καταρχάς, ευχαριστώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για, το, για την παρέμβαση που κάνετε για, τα, τα στατιστικά αυτά που έχετε. Θα κάνω ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Το σχόλιο ε, πρόκειται για το ότι είμαι ψυχίατρος στο επάγγελμα και όταν ασκούσα το επάγγελμά μου, πραγματικά τα στατιστικά στοιχεία για να τα βρει κάποιο ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Καλό είναι τα, να έχεις κάποιο οδηγό για να βρίσκεις τα στοιχεία, αλλά πρέπει η διαδικασία να απλοποιηθεί για το τελικό χρήστη και όχι μόνο για μεγάλους οργανισμούς. Αυτό είναι αναγκαίο γιατί πολλοί εκεί έξω κάνουμε δουλειά που τη χρειαζόμαστε άμεσα και όπως είπε και ο συνάδελφος ο Αντρέ, ε, χρειάζεται, είσαστε ένας μεγάλος οργανισμός. Μια, η ερώτησή μου είναι εξή. Συνεργάζεστε με 28 οργανισμούς που αποτελούνται από τα κάτι μελη Πώς εξασφαλίζετε, ποια κριτήρια βάζετε έτσι ώστε να πιστοποιείτε ότι τα στοιχεία που παίρνετε από αυτούς τους οργανισμούς είναι έγκυρα, αληθή και μπορούν να δημιουργήσουν μια προοπτική πολιτική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you. A very good question, which allows σας ευχαριστώ. Είναι πολύ καλό το ερώτημα σας και μου επιτρέπει να εξηγήσω το πώς λειτουργεί η στατιστική. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα γιατί αν δεν μπορούμε ε, να εξηγήσουμε γιατί τα δεδομένα μας είναι ακριβή, είναι ενημερωμένα και ούτω καθεξής, τότε δεν μπορούμε να τα παράσχουμε και να πείσουμε ότι πραγματικά μπορούν να εξυπηρετήσουν στην ενημερωμένη λήψη αποφάσεων. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα και υπάρχει ένας κανονισμός για τα στατιστικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει τις υποχρεώσεις της Eurostat και των κρατών μελών. Και να το πω ως αφήγημα. Δηλαδή, ξεκινώντα, θα πρέπει κανείς να διασφαλίσει ότι έχει συγκρίσιμα στατιστικά ε, στοιχεία, δηλαδή ε, τι ίδιε βάσει, τι ίδιε μεθοδολογίε. Και καταρχήν αυτό κάνουμε, δηλαδή συνεργαζόμαστε με τι υπηρεσίε έτσι ώστε να ακολουθούμε τι ίδιε μεθοδολογίε και να τι εφαρμόζουμε με τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε όλοι μα να ακολουθούμε τα ίδια πρότυπα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι τη εργασία που κάνουμε ω ε, Eurostat. Και αυτά τα πρότυπα τα οποία ακολουθούν όλοι οι μεθοδολογίε περιλαμβάνονται σε διαφορετικού κανονισμού. Μετά αρχίζουν και παράγονται τα δεδομένα από τι Εθνικέ Στατιστικέ Υπηρεσίε, μα αποστέλουν αυτά τα στοιχεία από την πλευρά του και εμεί έχουμε τα εργαλεία από δική μα πλευρά για να τα ελέγξουμε, ξεκινώντα από αμυγό αριθμητικά τεστ. Αν υπάρχουν δηλαδή ε, κάποιε αναντιστοιχίε μεταξύ των ίδιων των δεδομένων. Μετά κάνουμε και επιτόπιε επισκέψει στι διάφορε χώρε όπου ελέγχουμε δηλαδή τα βιβλία και στοιχεία, έχουμε και συγκεκριμένε διαδικασίε ελέγχου και από εκεί και μετά έχουμε και κάποιε διαδικασίε αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων, peer review. Όπου δηλαδή κάθε υπηρεσία θα πρέπει να εξηγήσει στις υπόλοιπες υπηρεσίες των άλλων κρατομελών πώς ακριβώς κάνουν τους υπολογισμούς για την παραγωγή των στοιχείων τους. Ε, και στη συνέχεια προβαίνουμε σε δημοσίευση ε, και ε, παρέχουμε και κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά για παράδειγμα δημοσιονομικά δεδομένα και ε, εκεί για παράδειγμα η Eurostat μπορεί να κάνει ένα σχόλιο λέγοντας ότι η Eurostat διατηρεί επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των λόγων δεδομένων και θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια μέτρα το, η αρμόδια υπηρεσία ούτω ώστε να αρθούν αυτές οι επιφυλάξεις της Eurostat. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές νομικές διατάξεις ανάλογα με το είδος των στατιστικών στοιχείων, γιατί ανά διαφορετικό πεδίο στατιστικών στοιχείων έχουμε διαφορετικό νομικό πλαίσιο κανονιστικό. Είναι λοιπόν και αυτό ένα κομμάτι, ακόμα και αν δεν γίνεται ορατό, τη δουλειά ε, που κάνει η ε, Γιώργο, Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που διασφαλίζει ακριβώ την ποιότητα ε, των στοιχείων. Ευχαριστούμε. Κυρία Γενική Διευθυντή, δεν θα παρατείνω την συζήτηση αυτή που ήταν ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα, αλλά έχουμε κάπω καθυστερήσει στην διάταξή μα Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την εξαιρετικά ενημερωτική, παιδαγωγική παρουσίασή σας και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όχι μόνο για τα νέα μέλη αλλά και για ιδιαίτερα απεπειραμένα μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό για εμάς να κατανοούμε τη σημασία που έχουν τα στατιστικά δεδομένα της δουλειάς ε, την οποία κάνει η Eurostat. Και πιστεύω ότι αυτή η ανταλλαγή μας επέτρεπε σε... να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα των στατιστικών δεδομένων στα πλαίσια της διαμόρφωσης των ε, πολιτικών μας σήμερα. Αλλά είναι σημαντικό διακύβευμα το, το θέμα της προ... της καταμέτρησης της ποσοτικοποίησης των προβλημάτων, ιδιαίτερα για τα κονδύλια που πιστώνονται στην κάθε προσπάθεια. Και, όπως και φυσικά οι δείκτες των επιδόσεων της κάθε παρέμβασης. Και πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα στοιχεία αυτά και να επικοινωνούμε διαρκώς. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με την ε, συνεδρία των συντονιστών το τμήμα της συζήτησης της, Επιτροπής, ε, της Επιτροπής ε, Ρέγγι τελειώνει εδώ. Σας ευχαριστώ και εγώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη για τα πολύ καλά ερωτήματά τους. Ε, πολύ χάρηκα αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να τα ξαναπούμε στην